Γεια σα, συνάδελφοι. Να αρχίσουμε γιατί όσοι έχουν πάρα πολλά θέματα και υποσχέθηκα όλου του εκλεκτού καλεσμένου ότι θα προλάβουν το αεροπλάνο του για να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή να τελειώσει η δουλειά του 16 και 40, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν καθένα τηρήσει ε, τα, τα, τα, τα, χρονικά όρια. Ε, έχουμε 18 γλώσσες ε, και δεν έχουμε κανένα έγγραφο, όλα είναι ηλεκτρονικά και μεταδίδεται και στο Ιντερνετ. Έχουμε επίση τα πρακτικά τη 26 Σεπτεμβρίου, τα οποία ε, υπάρχουν Ιντερνετικά, εκτό δεν έχετε κάποια σχόλια, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τώρα. Πάμε τώρα στην ακρόαση και καλώς όρισα οι εκπρόσωποι της ε, Fiat, ο κύριος Χάρολντ Western, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Χιάρε, Χιάρη μάλλον το πιο σωστό, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, παραγωγής και των ε, θεσμικών σχέσεων και ο κύριος Φωσάτη, ο οποίος είναι ο επικεφαλής σύμβουλος. Και τρεις θα λάβετε το λόγο κανονίστε μεταξύ ποιο θα λέει το λόγο, αλλά πρώτα θα μιλήσει ο κύριο Γουέστε. σα ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε και μέλη τη Επιτροπή. σα ευχαριστώ όλου για την ευκαιρία που μου δώσατε να συμμετάσχω σήμερα σε αυτή την ακρόαση και να σα παρουσιάσω τι ε, απόπειρε όσον αφορά τι εκπομπέ από του διζελοκινητήρε. Ε, ξεκινώ λέγοντα σας λίγα λόγια για, την, για τον όμιλο Fiat Chrysler. Είμαστε μια αυτοκινητοβιομηχανία, ένα όμιλο. Ε, αυτών των βιομηχανιών που σχεδιάζει, ε, τοποθετεί κινητήρες, κατασκευάζει και πολύ επιβατικά, ελαφρά εμπορικά και ε, επιχειρούμε σε περίπου 40 χώρες και επίσης έχουμε σχέσεις με πελάτες σε πάνω από 150 χώρες. Έχουμε πάνω από 230.000 εργαζομένους τους οποίους απασχολούμε. Και από την 31η Δεκεμβρίου του 2015 έχουμε 164 κέντρα και εγκαταστάσεις και αυτό καλύπτει και τα, επι, τα επιβατικά, τα ελαφρά εμπορικά και επίση ε, τι εγκαταστάσει για τα ανταλλακτικά. 40 στην Ιταλία, 35 στην υπόλοιπη Ευρώπη, 29 στη ΣΥΠΑ, 22 στην Βραζιλία, 14 στο Μεξικό και 6 στον Καναδά και οι υπόλοιπε εγκαταστάσει και εργοστάσια στην Αργεντινή, την Κίνα και σε άλλε χώρε. Το 2015 ο Όμιλος ε, είχε πωλήσει ε, πάνω από 4,6 εκατομμύρια επιβατικά και ελαφρά εμπορικά οχήματα. Από αυτά πάνω από το 1 εκατομμύριο ε, πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος επίσης έχει αξιόλογη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης. Από τον Δεκέμβριο του 2015 έχουμε ερευνητικά κέντρα τον αριθμό 84 σε όλο τον ε, κόσμο και απασχολούμε εκεί περίπου 20.000 ε, πρόσωπα. Αυτή είναι ειδική σε πολλούς κλάδους, ε, είναι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, μηχανικοί, υλικά, επίση και στην πληροφορική. Το 2015 το 2015 οι δαπάνες μας όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη ήταν περίπου 4 δισεκατομμύρια, δηλαδή 3,6% των καθαρών εσόδων από την δραστηριότητα τη βιομηχανική. Αυτό σήμερα ότι είχαμε 14,5 το 2014 και ε, επίσης αυτό σημαίνει ότι ήμασταν στο 7,6% ως αύξηση από τα 3,2 δις που ήταν το άθροισμα αυτών των ε, εσόδων το 2013. Οι ποιε δραστηριότητε ε, τώρα επικεντρώνονται τα εξή. Πώ θα μειώσουμε τη βλάβη στο περιβάλλον από τα οχήματά μα, πώ θα μειώσουμε τον θόρυβο, το διοξίδιο του άνθρακα και τα άλλα ρηπαντικά. Επίση, πώ θα είναι πιο αποτελεσματικά τα όργανα, συγγνώμη, τα, τα οχήματα και πώς θα μπορούμε να έχουμε την ανάκτηση και ανακύκλωση όταν κλείσουν τον κύκλο τους. Να ε, έχουν περισσότερη ασφάλεια, ενεργειακή, ενεργητική, παθητική και επίσης να μπορούμε να έχουμε οχήματα τα οποία να είναι ευφυή και να πιάνει και τόπο η πληροφορική και θέλουμε επίσης να έχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα, καινούργια αρχιτεκτονική ούτως υπήν, ε, απόδοση, άνεση και καινοτομία και ταυτόχρονα οικονομική βιωσιμότητα όσον αφορά την των οχημάτων. Και τώρα βλέπουμε ότι έχουμε τεχνογνωσία και έρευνα σε πάρα πολλούς ε, κλάδους της μηχανία και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως ε, ε, το νομοθετικό, το κανονιστικό περιβάλλον μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 70 διαφορετικούς κανονισμούς οι οποίοι καλύπτουν αυτή την έγκριση τύπου όσον αφορά τη διαδικασία προέγγισης αυτοκινήτων και ο όμιλός μας έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις τεχνολογίες για τους κινητήρες αλλά και να έχουμε εναλλακτικά συστήματα κίνησης. Και στο τελευταίο μας business plan επαναλάβαμε την δέσμευσή μας όσον αφορά το να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τεχνολογίες ε, για ηλεκτρική κίνηση κίνηση και να έχουμε πολλές εφαρμογές όπως και οχήματα που να λειτουργούν με μπαταρία, τα υβριδικά πρώτης γενιάς με, με σημαντικούς κινητήρες και αυτά που είναι μόνο με ρεύμα από την ε, μπρίζα. Ε, επίσης, Επίση, μπορέσαμε να επενδύσουμε σε κάποια πάρα πολύ καθαρά καύσιμα ότι υπάρχει σήμερα φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, βιομεθάνιο και προσφέρουμε τεχνολογίε οι οποίε βοηθούν τόσο ώστε να είναι πιο λίγε εκπομπέ όσον αφορά τα καύσιμα που υπάρχουν κάστοτε και σε κάθε αγορά. Εμεί ξεκινήσαμε την ανάπτυξη κινητήρων από φυσικό αέριο αρχή τη δεκαετία του 90 και από τότε είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά αυτή την αγορά στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα 12 μοντέλα επιβατηγών και ελαφρών εμπορικών και πουλήσαν το 2015 πάνω από 44.000 οχήματα, το οποίο σημαίνει το 50% της ευρωπαϊκής αγοράς. Από το 1997 δε ο όμιλός μας έχει πουλήσει πάνω από 700.000 οχήματα ε, τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο. Σήμερα όμως αυτό που είναι το θέμα μας είναι οι εκπομπές από τους πρωτα Πρώτα-πρώτα, για ποιο λόγο έχει αυξηθεί η αγορά των διζελοκινήτων στην Ευρώπη. Η τιμή του δίζελ ε, ιστορικά είναι κάτω από την τιμή της ε, βενζίνης ακόμα και τώρα κατά μέσο όρο 10% πιο φτηνό είναι το ντίζελ και κατανάλωση 20-25% πιο κάτω από την κατανάλωση των ε, βενζινοκινητήρων. Και επίσης υπάρχουν ε, επιδόσεις, υπάρχει αξιοπιστία αυτών των κινητήρων και αυτό το, ε, εκτιμούν οι ιδιοκτήτε των αυτοκινήτων πάση κατηγορία και ιδίω εκείνοι που κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Δεν θα ήταν δε δυνατόν να μπορέσουμε να ε, τηρήσουμε του στόχου, του φιλόδοξου τη μείωση των εκπομπών του δεξιδίου 95 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο το 2021 χωρί να υπάρχει η τεχνολογία του διζελοκινητήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα επιβατικά αυτοκίνητα με διζελοκινητήρα τώρα αντιπροσωπεύουν το 50% τη αγορά. Όσον αφορά δε την, τον όμιλό μας αυτό το νούμερο σημαίνει 38% κάπως λιγότερο. Τώρα όσον αφορά τα ελαφρά ε, εμπορικά ε, είναι γνωστό ότι η αγορά καλύπτεται σχεδόν 100% από τις ελοκινητήρες. Από πλευράς τώρα τεχνικής, η κατασκευή της ελοκινητήρων που να συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές της κατηγορίας Euro 5 σημαίνει το εξή. Σε δύο μέτωπα έπρεπε να κατευθυνθούμε. Πώς θα μειωθούν οι εκπομπές ε, κατά την συμπίωση, αυτό που ονομάζουμε EGR ε, και επίσης θα έπρεπε να γίνει μια επεξεργασία των ρηπαντών πριν την εκπομπή μέσω του καταλήτη. Αυτό που λέμε DOC, Diesel Oxidation Catalyst. Και να υπάρχει και αυτό το φίλτρο των μορίων σωματιδίων και στη συνέχεια πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις εκπομπές της κατηγορίας Euro 6B. Οπότε ο όμιλός μας προσέθεσε το, e, το SCR, Selective Catalytic Reduction, μια τεχνολογία για κάποια μοντέλα που έχουν υψηλότερη ενεργειακή απέτηση. Και είχαμε επίσης τον καταλήτη για τον NOx, για, το, για τα οξύδια του αζότου του χρόνου. Θα έχουμε καινούργιες ε, ε, ε, διαδικασίες για τα τεστ, δοκιμές, για να μετρήσουμε τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, RDE, και επίσης θα, δούμε τι θα γίνει με τους νέους κανόνες ε, και την καινούργια διαδικασία WLTP για τα ελαφρά εμπορικά. επίσης, έτσι θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και οι καταναλωτές και η βιομηχανία. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη αυτών των αλλαγών Τη Δευτέρα Φεβρουαρίου τρέχοντος έτου ανακοινώσαμε ω όμιλο ότι θα αναβαθμίσουμε ε, το, τα τεστ και ότι εκουσίως πρόκειται να αναβαθμίσουμε ε, την προσαρμογή του μας όσον αφορά το Euro 6B με καινούρια δεδομένα, με καινούριο λογισμικό, ούτω ώστε να έχουμε καλύτερε επιδόσει όσον αφορά τι εκπομπέ σε πραγματικέ νίκε οδήγηση. Και αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά όλου του τζενοκυλητήρε μα που παράγονται. Και ε, αυτού του είδους η αναβάθμιση του λογισμικού έγινε δωρεάν προς όλους τους ιδιοκτήτες ε, όσων αυτοκινήτων έχουν τέτοιου διζελοκινητήρες ε, και ε, φέτος θα ολοκληρωθεί αυτό. Τέλος, εφαρμόζουμε αυτή τη νέα δικασία RD και θα έχουμε το SCR επίσης, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει ένα κόστος, παραπάνω κόστος. Και ίσως αυτό ίσως δεν είναι βιώσιμο όσον αφορά τις ελοκινητήρες για πολλά από τα πιο φτηνά μας μοντέλα. Πριν φτάσουμε στην ώρα των ερωταπαντήσεων θα πρέπει να σας πω και κάτι τελευταίο. Ως γνωρίζετε, στη Γερμανία η KBA διαφωνεί με κάποια στοιχεία όσον αφορά ε, τις απόψεις της ε, Ιταλικής αρχής που ασχολείται με την έγκριση τύπου για τα οχήματα Euro 6. Αυτό οδήγησε σε διαμεσολάβηση και αυτή βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη. Ε, όσο λοιπόν έχουμε αυτού του την εκκρεμωδικία δεν θα πρέπει εμείς να συζητήσουμε ό,τι καλύπτει αυτού του είδους η διαμεσολάβηση, αυτή η διαιτησία που θα την πούμε, ε, είναι θέμα εμπιστευτικότητα και, και για τους προμηθευτές. Οπότε σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για αυτό. Ε, ό,τι λοιπόν δεν μπορούμε να απαντήσουμε, ευχαριστώ που καταλαβαίνετε γιατί πέραν αυτού, περιμένω τις ερωτήσεις σας για να μπορέσω να σας παράσχω ό,τι θέλετε ως ε, στοιχεία και πληροφορίες. Ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Βέστα. Ε, βέβαια, γίνονται ερωτήσεις γενικές, έτσι. Ε, ελπίζουμε να μπορέσετε να απαντήσετε όσο γίνεται περισσότερες. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ο κύριος Γκερμπράντη πρώτος. Madam thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Βέστερ και για τις γραπτές σας απαντήσεις και για τη σημερινή σας τοποθέτηση. Πρώτη ερώτηση αφορά την απάντηση ε, στην ερώτηση 2 για τους μηχανισμούς εξαπάτησης. Και λέτε ε, ότι ε, δεν καλύπτεται από τις εξαιρεσει ένα σύστημα το οποίο βλέπει ότι γίνεται δοκιμή εκείνη την ώρα και το εξαπατά. Δηλαδή επικεντρώνεστε μόνο σε εκείνε τι σύσκευέ ή ε, το λογισμικό που δείχνει ποιο είναι το αυτοκίνητο που γίνεται ή, το λογισμικό που δείχνει ποιο είναι το αυτοκίνητο που γίνεται η δοκιμή αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αυτό αφορά οποιοδήποτε στοιχείο και με διάφορα χαρακτηριστικά που μετράνε ή διάφορες άλλες παραμέτρους ε, με στόχο να ενεργοποιήσει, να ε, αλλοιώσει, που μιλάμε για τη ΦΙΑΤ, να καθυστερήσει ή να απενεργοποιήσει ε, τον έλεγχο κτλ. κτλ. Άρα, έχω την αίσθηση ότι χρησιμοποιείται ένα πάρα πολύ περιορισμένο ορισμό ε, της συσκευή μηχανισμού εξαπάτησης σε σχέση με την αρχική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. I would like to go back to 2007 2008 when the was born. Θα ήθελα να επανέλθω στο 2007 και 2008. Ξέρετε ότι στο 310, άρθρο 310, ακριβώς γράφει αυτά που είπατε κι εσείς. Εγώ προσωπικά πιστεύω και το ερμηνεύω έτσι, ότι ήταν γνωστό, εξακολουθεί να είναι γνωστό και είναι απαραίτητο, ε, τα άρθρα 5, 1 και 2 και λένε το 1. Ο κατασκευαστής θα φροντίζει ο εξοπλισμός με τρόπο ώστε να κατασκευάζονται και να εργολογούνται τα οχήματα με τρόπο ώστε να μπορούν να μορφώνονται με την νομοθεσία και τα εκτελεστικά μέτρα για τις εκπομπές. Η χρήση των defeat devices μειώνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου εκπομπών. Ε, θα απαγορεύεται. Η απαγόρευση δεν θα εφαρμόζεται όταν αιτιολογείται η ανάγκη για να προστατευτεί ο κινητήρας ε, κατά τη ζημιάς ήταν ατυχημάτων για να λειτουργεί με ασφάλεια το όχημα. Δεύτερον, η συσκευή δεν υπερβαίνει τις απαιτήσει ε, της έναρξης ε, του, του κινητήρα και επίσης ε, κατά τη διαδικασία δοκιμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εξατμίσεις, δηλαδή τι εννοούμε. Στην πρώτη περίπτωση απαγορεύεται το defeat ε, στη δεύτερη περίπτωση, μέσα στο λογισμικό, τίποτα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι το όχημα ε, συμμετέχει σε μία δοκιμή. Ο κύριος Γκεμπράντη, ναι, αλλά με αυτόν τον ορισμό που διάβασα εγώ, αυτό το τελευταίο τμήμα του ορισμού σας δεν έχει σχέση, δεν λέει ότι είναι defeat devices όταν αναγνωρίζει τη δοκιμή το όχημα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν βλέπω να, το χρονόμετρο Πρόεδρος, ναι, έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Άλλο 1,5 λεπτό έχετε, κύριε Γκυμπράντη. Μπορώ κι εγώ να, ε, χρησιμοποιώ τέτοια τυφή devices για το χρόνο. Ε, λοιπόν, όπως προκύπτει από τις 2 Φεβρουαρίου, του τρέχοντος και από ό,τι είπατε, ε, ε είναι, σύμ, από όσο το παρουσιάζετε εσείς φαίνεται να είναι σύμπτωση λίγους μήνες μετά το Σεπτέμβρη, γίνεται να κάνετε εσείς τεχνικές ρυθμίσεις ώστε ε, να μην προκαλεί ζημιά στο κινητήρα η τεχνολογία μείωση των εκπομπών και άρα να μην χρειάζεται είτε να διακοπεί η λειτουργία της είτε να ρυθμιστεί αλλιώ τεχνικά. Μπορείτε να με εξηγήσετε γιατί τώρα είναι δυνατό και όχι όταν κατασκευάστηκαν και ετέθηκαν στην αγορά αυτά τα οχήματα. Εγώ κατάλαβα ότι είναι επικαιροποίηση λογισμικού. Γιατί ο κινητήρα. ε, ε, προκαλεί το ζημιά στο κινητήρα τότε και ξαφνικά τώρα με το update του, του Φεβρουαρίου και την αλλαγή του λογισμικού δεν ε, ε, προκαλείται ζημιά στο κινητήρα. Εφού δεν έχουμε χρόνο, δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και να σας περιγράψω όλα τα θέματα που έχουμε με τους κινητήρες. Ε, όλοι κάνουν πολλές δοκιμές και εμείς φυσικά εκατομμύρια χιλιόμετρα και εκατομμύρια επικατομμυρίων για κάθε νέα τύπο και μοντέλο και ε, κάθε χιλιάδες ωρών δοκιμές σε δικαστήριο. Για να κάνεις ένα ε, καινούριο καλυβράς χρειάζεσαι 12 με 14 μήνες. Και αρχίσαμε τέλη του 2014, συνεχίσαμε το 2015 και αυτό δεν συνδεόταν με το θέμα που ενέκυψε το Σεπτέμβριο. Κάναμε 16.000 ε, ώρες δοκιμές ε, ε, εργαστηρίου, πάνω από 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα και δεκάδες χήματα. Γιατί το κάναμε αυτό όμως. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, το 2012 νομίζω, εισήχθη ένα σύστημα και τα επόμενα χρόνια ε, κάναμε αναβαθμίσει. αυτό λέγεται eco drive. Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω και πάλι ο κύριο Γκεμπράντη. Έτσι ε, θα μακρηγορήσουμε και θα πλατιάσουμε και θα χάσουμε χρόνο. Όπως λέτε εδώ και καιρό το σχεδιάζετε και τώρα μπορέσετε να το κάνετε. Τώρα, γιατί χρησιμοποιήσετε τεχνολογία που μειώνει τι εκπομπέ ε, και δεν μπορεί να ανάψει σε κανονική χρήση σε κανονική χρήση χωρίς να βλάψουν τον κινητήρα σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω επίση γιατί τον έκριναν αυτό οι Ιταλικέ αρχέ. Δική σα είναι η τεχνολογία που μπορεί να ε, προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα. Οι ανταγωνιστέ σα χρησιμοποιούν μια τεχνολογία που δεν ε, βλάπτει του κινητήρε. Γιατί το δέχτηκαν αυτό τον έκριναν. Πρώτον, εμείς ούτε ανάβουμε ούτε σβήνουμε, τροποποιούμε. Υπάρχουν νόμοι και κανονισμοί και αυτό που πριτανεύει πάντα είναι η ασφάλεια και για τον οδηγό. Πάνω από 100.000 ε, πελάτες μας αγοράζουν κινητήρες Euro 6 και μας αναφέρουν λεπτομερώς πώς χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα και αυτό μας βοήθησε να ξανακάνουμε τις προσαρμογές μας ε, και να επαναπροσδιορίσουμε τους κινδύνους. Ο κύριος Άλμπα. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ρωτήσω κάτι για τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις εκπομπές ε, καυσαέριων. Μ' ακούτε? No. I Ναι, έχω διερμηνία, εντάξει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι για την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως απόκριση στο σκάνδαλο και θέλω και την εκτίμησή σας. Πιστεύετε ότι με αυτή τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέλλον θα αποτρέπονται τέτοιου είδους σκάνδαλα και επίσης πιστεύετε ότι με αυτή την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πετρελαιοκίνηση είναι ασφαλής και βιώσιμη επιλογή για το μέλλον και οι εργαζόμενοι ε, σε αυτό το κλάδο στην αυτοκίνητο βιομηχανία που παράγει αυτοκίνητα δίζελ θα έχουν δουλειά, είναι βιώσιμος αυτός ο κλάδος και κερδοφόρος όπως σας είπα. Ο μόνος τρόπος να προσαρμοστεί κανείς και να συμμορφωθεί ε, με τον νέο κύκλο έρευνας και ανάπτυξης είναι ο ε, ενεργός κινητήρας SCR e real, uh, driving um, conditions. Hmm. Έχει ως εξής, δηλαδή, θα πρέπει να είναι δύο προς ένα η κατανάλωση ε, πετρελαίου σε σχέση για, την εκπομπή ε, λοιπόν ρήπων και μεταξύ αυτών. Ε, τώρα έχουμε 80 γραμμάρια στο χιλιόμετρο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σε μια συμμόρφωση με αυτά τα όρια. Ε, Μάλιστα. Και εσείς πιστεύετε ότι η προσαρμογή συγκεκριμένων γιοταχή που κινούνται με δίζελ με επιπλέον τεχνολογία περιορισμού των καυσαερίων είναι βιώσιμη ε, λύση και εναλλακτική. Μάλιστα. Το πιστεύω. Και όπως σας είπα, έχει σημασία για όλους τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και στην Ευρώπη που είναι τόσο πολλά τα πετρελοκίνητα και Όσο ανεβαίνει ο αριθμό των αυτοκινήτων, τόσο πιο σημαντικό είναι. Θα πρέπει να παραμείνουν τα πετρελοκίνητα ε, στο στόλο των ε, οχημάτων που κυκλοφορούν, γιατί υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ο κύριο Γκίζικε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους κυρίους της ΦΙΑΤ που ήρθαν σήμερα στην Επιτροπή μας, ο κ. Βέστερ, ο Ροζάτη, κύριε Κιάρη. Κύριε Βέστερ και γερμανικά καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεστε ε, μετάφραση, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Στην εισαγωγική σας παρουσίαση ε, είχατε μία αίρεση, ένα περιορισμό για τη διαδικασία ε, συνδιαλλαγής του γερμανικού οργανισμού έγκρισης με τον Ιταλικό μπορείτε να μου απαντήσετε στην εξή ερώτηση. Αν καταλήξει ο γερμανικός οργανισμός ότι είναι παράνομο μετά από 22 λεπτά να διακόπτεται ε, αυτό το σύστημα, τι θα κάνετε, ε, δεν θα εισάγουμε από την Ιταλία αυτοκίνητα. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Μετά τις δημοσιεύσεις ε, του οργανισμού αυτού, του γερμανικού, έχει ανακρούσει πρίμνα. Σήμερα τι λένε, ότι το σύστημα καθαρισμού ή επεξεργασίας των καυσαερίων μετά από 22 λεπτά ε, ε, έχει κάνει κάποιες μετρήσεις. Ζητώ συγγνώμη τώρα που θα πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Έχει μετρήσει ο γερμανικός Οργανισμό η Ομοσπονδία Υπηρεσία, ε, υπηρεσία Αρχημάτων, τα συστήματα υψηλής και χαμηλής πίεσης στις βαλβίδες, ε, που δεν είναι γραμμικά συστήματα, είναι σε μεγάλο βαθμό. Μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, ε, ότι αν ανοίξετε μία βαλβίδα, δεν ρέει έτσι με αναλογικό τρόπο πάντα ναι, πολύ τεχνικά μας τα λέτε αυτά, αλλά δεν καταλαβαίνω. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Εγώ τεχνικά δεν σκαμπάζω. Τι σημαίνει modulation μετά από 22 ε, λεπτά. Τι τροποποιείται. Περιορίζεται η αποτελεσματικότητα και αν ναι, ε, ποσοστία πώς το μετράτε αυτό και σε ποια τάξη μεγέθους βρίσκεται. Αυτό σημαίνει η τροποποίηση, η μετριασμός των συστημάτων ε, καθαρισμού των καυσαερίων ότι πρώτον το μείγμα υψηλής πίεσης και χαμηλής πίεσης ε, για την επιστροφή των καυσαρίων πρέπει να αλλάξει. Ε, ε, έχει να κάνει αυτό με τη θερμοκρασία, με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και με την απόδοση επίδοση του αυτοκινήτου. Και μετά πρέπει να αλλάξει και το DNOx που έχει να κάνει με τα οξύδια του αζότου. Και μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Στις γραπτές σας απαντήσεις για την ερώτηση 2 λέτε ότι δεν υπάρχει όχημα diesel που να περνάει τον έλεγχο της εντατικής χρήσης. Έχουμε 20 λεπτά ε, στο εργαστήριο. Υπάρχει μια διέρεξη με τη δική σας εταιρεία για τα 22 λεπτά. Από πότε θα πρέπει στη Fiat και μετά να, να σβήνει αυτό το σύστημα. Μα πόσες φορές πρέπει να το πω ακόμα. Δεν σβήνουμε τίποτα. Δεν σβήνουμε δεν απενεργοποιούμε τίποτα. Καλά, στη ε, συνέχεια θα τα πείτε εσείς. Ε, ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε λεπτομέρειες. Αυτό εξαρτάται από το αυτοκίνητο, από πάρα πολλούς παράγοντες και παραμέτρους. Καλώς, ε, Πρόεδρος. Η κυρία ε, Βονταλόν. Ευχαριστώ, θα μιλήσω γαλλικά. Okay. Okay. Merci. Euh, bon, je vais pas vous parler, euh, δεν θα σας μιλήσω για τα 22 λεπτά γιατί σας έθεσαν αυτό το ερώτημα. Θέλω να μιλήσω για άλλες δοκιμές που έγιναν. Στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα είχαμε την Ούτα Ξεράμε και μας μίλησε για το ΦΙΑ το 500 που δοκιμάστηκε και έγιναν τρεις διαφορετικές δοκιμές όπως καλά ξέρετε. με 11.500 χιλιόμετρα και RGE Plus ε, σύστημα καθαρισμού 68,2 mg το χιλιόμετρο για τα NOx η πρώτη δοκιμή ε, σε εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι φτάσαμε στα 246,7 mg το χιλιόμετρο το D2 με ζεστό κινητήρα 528,5 ε, ε, μιλιγκράμμ το χιλιόμετρο και στην πίστα εκτός εργαστηρίου δηλαδή, όχι ένα λεπτό, το D2 όχι, το είπα αυτό. Και το D3, 1354 ε, μιλιγκράμμ το χιλιόμετρο. Μπορείτε να εξηγήσετε αυτές τις διαφορές. Υπήρξε πρόβλημα με το καθαρισμό των ρήπων. Γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην έγκριση τύπου και τα αποτελέσματα που είχαμε από την Επιτροπή Ελέγχου. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω όλα αυτά τα αποτελέσματα δοκιμών. Μόνο μπορώ να σας πω ότι είναι καλές οι επιδόσεις των οχημάτων μας. Είμαστε, έχουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία. Από πέρσι το Σεπτέμβριο γίνονται πάρα πολλές δοκιμές παγκοσμίω από διάφορους ε, οργανισμούς και χρησιμοποιούνται διαφορετικές μεθοδολογίες. Την Παρασκευή το βράζει. Είδα κάτι που μια δοκιμή του Ολλανδικού Ινστιτούτου πήρε ένα Grand Cherokee και τα στοιχεία, τα αποτελέσματα καμία σχέση δεν είχαν ε, με τα αποτελέσματα τα δικά μας. Ε, ε είχε 150 χιλιόμετρα στο κοντέρ. Ζητώ συγγνώμη που μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Διακόπτη η κυρία Νταλόν Μπονφουά. Ζητώ συγγνώμη, δεν μιλάμε με, ε, για 150.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα είχε το αυτοκίνητο. Απλώς ε, είναι χάσμα ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία της έγκρισης τύπου και των δοκιμών. Το πρώτο ήταν και σε εργαστήριο το τεστ. Καταλαβαίνω ότι μπορείτε να αμφισβήσετε μετρήσεις που έχουν γίνει αφήσιμους οργανισμού σε διάφορα κράτη-μέλη. Δεν μπορείτε όμω να αμφισβητήσετε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τον ε, καθαρισμό των ρήπων. Το πρώτο σύστημα προτείνεται. Απάντηση. Δεν έχω εξήγηση να σα δώσω για, για αυτές τις το είπα. Αυτές οι τιμές δεν θα έπρεπε να παρουσιάζουν τέτοιες διαφορές. Δεν έχω ενημέρωση για τις δοκιμές, για τις συνθήκες της δοκιμής, για την κατάσταση των αυτοκινήτων. Αυτό που ξέρουμε, και αυτό ισχύει και για το διοξίδιο του άνθρακα, ισχύει και για τις εκπομπές που συζητάμε εδώ, είναι ότι ο Ευρωπαϊκός κύκλος δοκιμών που άρχισε από την αρχή της δεκαετίας του 1970 και συνεχίζει και μέχρι σήμερα, μετράμε εκπομπές υπό προκαθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες. Αυτά τα αποτελέσματα λοιπόν δεν μπορούν από επιχειρησιακής, από λειτουργικής πλευράς να ε, είναι εγγυημένα. Για κανένα όχημα. Ναι, βεβαίως δεν μπορείτε να το εγγυηθείτε. Αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στα ε, φυσικά θα υπάρχουν παρεκκλήσεις και διαφορές. Ε, είναι πολύ μεγάλη η στρέβλωση και καταλαβαίνετε και τους καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν το όχημα και η πραγματικότητα είναι 300-400 φορές υψηλότερη από τις ε, τιμές των εργαστηρίων. Το να αυτό. Απάντηση. Ε, μόνο στη στοιχεία συγκρίσιμα μπορώ να σχολιάσω. Αν το σβήσετε, σβήσετε όλα τα συστήματα ελέγχου εκπομπών, δεν, δεν, αυτό δεν είναι τεχνική ρύθμιση, είναι απενεργοποίηση. Οπότε δεν μπορείτε να μπείτε στην κατηγορία 12. Κύριε Χέγκελ. Γεια σας κύριε Βέστα. Έχω την εξής ερώτηση, την οποία πανελειμμένα έχω κάνει και σε εσά. Πιστεύετε ότι οι αρχικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν υπερβολικά ασαφείς. Δεν μιλώ για τη fit devices, Θα εξηγήσατε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται συστήματα εξαπάτησης, αλλά μήπως ήταν υπερβολικά όριστα και ασαφή ε, ε, όσα ίσια και όλα αυτά που συζητούνται πέρα από τα defeat devices ε, συνδέονται με τα προηγούμενα. Συμφωνώ απολύτως κύριε Χένκελ. Για ποιο λόγο. Ε, διότι θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Από την αρχή της δεκαετίας του 70 έχουμε εφαρμόσει όλοι τις προδιαγραφές NEDC για τις δοκιμές και θεωρούσαμε όλοι, ήμασταν ε, πεπισμένοι ότι αυτός ο κύκλος δοκιμών ανταποκρίνεται, εκεί θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει μια κανονική χρήση οχημάτων. Σήμερα δεν ισχύει πια αυτό. Α, αυτό. Και δεύτερον, εμείς είμαστε ένας όμιλος Το μισό καιρό μου το βερνάω περίπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τον Αμερικανικό ε, ε, οργανισμό, ΕΠΑ κλπ. Χωρίς να θέλω να σε λεπτομέρειες, βασική διαφορά της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής με κινητωμένων πολιτιών για αυτά τα θέματα ποια είναι. Ότι οι νόμοι έχουν ε, σωστή σύλληψη και σκέψη από την κατασκευή τους. Ε, είναι πάρα πολύ λεπτομερής και στην νομοθεσία και στις εκτελεστικές και στις εφαρμοστικές διατάξεις. Είναι πάρα πολύ πιο αυστηρή και πάρα πολύ πιο ακριβής από ό,τι ήμασταν εμείς μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Άρα και ε, σε συνδυασμό με νέους κύκλους για real drive emissions, για εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και μέτρησή τους θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό και πολύ συγκεκριμένα να περιγράψουμε ε, τι θέλουμε και τι περιμένουμε από αυτά τα συστήματα στην καθημερινή κανονική οδήγηση. Θα θεωρούσατε σκόπιμο, κύριε Βέστε, οι οδηγίε για τα καυσαέρια στην Ευρώπη και στην Αμερική να προσαρμοστούν, να συμπλιάσουν, να εναρμονιστούν. Για μας θα ήταν θαυμάσιο αυτό και ε, σπουδαία βοήθεια. Ε, γιατί αποκλίνουν οι οδηγίε όχι μόνο για τα καυσαέρια και έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτά, αλλά και για άλλα θέματα. Είναι πολύ μεγάλο κόστος. Παράδειγμα, όταν το Fiat το 500 πήγε στην Αμερική, πώς να το πω, έπρεπε να αλλάξουμε τελείως οι ελοκαθαριστήρες, διότι οι Αμερικανοί έχουν διαφορετική ε, διάταξη για τους ελοκαθαριστήρες αλλά δεν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν έξω από το τζάμι, γιατί να τους αλλάζαμε. Στις διαπραγματεύσεις για το TTIP πιστεύετε ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί. Ναι, θα το καλωσορίζαμε κάτι τέτοιο, θα το ευχόμασταν. Για το Diesel βεβαίως θα πρέπει το κέντρο βάρους να είναι στην ευρωπαϊκή πλευρά, διότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίζηση δίζελ για γιοταχή και ελαφρά επαγγελματικά είναι 3% ενώ εμάς περίπου 50% είναι στα γιοταχή και περίπου 100% στα επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, είπατε απαντώντας σε άλλη ερώτηση ότι οι αμερικανικές προδιαγραφές είναι τόσο πιο, ε, σαφέστερες και ακριβέστερες και τα λοιπά και, και πιο απαιτητικέ δεν θα είχε νόημα να προσαρμοστούμε κι εμείς και να συμμορφωθούμε σε αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε τόσους πολλούς πετρελοκινητήρες. Μήπως θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε και προσανατολιστούμε περισσότερο στις αμερικανικές προδιαγραφές. Ναι, αλλά αν συμφωνήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί του άνθρακα, γιατί δεν ξέρω καμία τεχνολογία που να το αντισταθμίζει αυτό. Πριν από μια εβδομάδα είχε έρθει ο κύριο Σεράριο από το ε, Ιταλικό Υπουργείο Συγκοινωνιών και Μεταφορών και μας είπε ότι στη Fiat δεν υπάρχει σύστημα εξαπάτησης, defeat device, αυτό που είπατε κι εσείς. Και αυτό που το ξέρει. Μα έχουν γίνει δοκιμέ. Δοκιμέ, τι δοκιμέ έχουν. Τι έγινε, έκανε δοκιμές στο Υπουργείο Μεταφορών τη Ιταλία και το ξέρει. Ναι, βεβαίω. Υπάρχει το θέμα witness testing, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο ευρύτατα, όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και όπως γνωρίζετε αυτό σημαίνει ότι επειδή το κόστος είναι τεράστιο και αυξάνεται όλο και περισσότερο για τέτοιου είδους δοκιμές, είναι πάρα πολύ σοφιστική και περίπλοκα τα συστήματα αυτά. Και για την έγκριση τύπου παντού στον κόσμο και στις ΗΠΑ και στην Κίνα γίνονται οι δοκιμέ παρουσία πολλές φορές του οργανισμού που δίνει την έγκριση που Πάνε ε, στα εργαστήρια και είναι παρόντες βεβαίω και τα Υπουργεία. Κύριο Πέντερλε. Σα ευχαριστώ πολύ. Μας εξηγείτε ότι δεν χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα παράκαμψης. Αυτό γίνεται και στα οχήματα που πουλάτε στις ίπα. Ε, Άρα παρακάμπτεται τους ελέγχους και την νομοθεσία. Ακόμα και όταν δεν λειτουργεί αυτή η πλακέτα, αυτό το σύστημα. Όχι, όχι, δεν κλείνω ποτέ. Δεν είναι ποτέ off. Λέει ο κύριος από τη Fiat. Πόσα αυτοκίνητα diesel πουλάτε στη ΣΥΠΑ. Σας είπα όχι τόσα πολλά. Μόνο 3% στις ε, είπα είναι οι κινητέ. Πολύ, πολύ χαμηλό όπως είπαμε. Ε, μίλησα πριν για 20.000 ετησίως. Περισσότερα στον Καναδά και λιγότερο ε, αυτά αφορούν τη ΣΥΠΑ. Οπότε υπάρχουν οι ορικές τιμές από την νομοθεσία. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε αυτό. Τι θεωρείτε πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε προ τη νομοθεσία, να περάσετε τις δοκιμές και να εξασφαλίσετε ότι όταν κανείς πραγματικά οδηγεί τηρούνται αυτέ οι ωραϊκέ τιμέ. Βέστερ. Δεν υπάρχει λεπτομεριακή νομοθετική ρύθμιση. Η ΦΙΤ έχει συμμετάσχει σε κάποιες ομάδε εργασία γιατί από ό,τι ξέρω πολλοί, πολλοί όμιλοι αυτοκινητοβιομηχανών έχουν συμμετάσχει, αλλά η Fiat έχει ποτέ συμμετάσχει. Western. Ναι, έχουμε συμμετάσχει όπως και οι άλλες ε, βιομηχανίες μέσω της ΑΣΕΑ και έχουμε συζητήσει τα σχετικά. Άρα θεωρείτε ότι ορθώς έχει ερμηνευτεί ο νόμος. Όπως έχουμε σήμερα τα πράγματα του κύριου Βέστερ, άφορ τον φορέα των αυτού και των ε, ρυθμιστικών αρχών απ' την άλλη. Δεν με καλύπτει αυτό που απαντήσατε, γιατί σε πολλές από αυτές τις ομάδες ε, εργασίας έχουμε πολλούς εκπροσώπους της βιομηχανίας. Έτσι θεωρούμε ότι είναι το σωστό να γίνει. Να μην πέταμε στο παιχνίδι τη βιομηχανία, αλλά ε, να υπάρχουν οριακές τιμές οι οποίες να είναι ρεαλιστικές. Στην Ευρώπη θεωρούμε ότι έχουμε πιο ψηλά στάνταρα από τον υπόλοιπο κόσμο. Όμως πολλές φορές έχουν πολύ πιο απαιτητικά στάνταρα στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα τι γίνεται με αυτές τις ομάδες εργασίας και την ομοθεσία; Βέστερ, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να νομοθετήσει ε, αφήνοντας απ' έξω την βιομηχανία γιατί εμείς έχουμε όλη την τεχνογνωσία. Και στην αρχή, αρχή σας διάβασα τα άρθρα 5,1 και 5,2, τις δύο αυτές παραγράφους. Και είχαμε συμμετάσχει σε αυτές τις ομάδες στο δεύτερο μισό από το 2005-2010 και εγώ από ό,τι κατάλαβα Πρώτον ήταν κατηγορηματική η διάταξη που αφορούσε αυτές τις συσκευέ παράκαμψης, όπως και να τις λέγανε. Και κατόπιν ονομάζουν κατονομάζονται, αναφέρονται κάποιες εξαιρέσεις. Από τη μία μεριά η βιομηχανία, από την άλλη οι ρυθμιστικές αρχές. Δεν θα κάνανε αυτή τη συνάντηση, αν δεν ήταν αναγκαίο, να πιέσει τώρα ο χρόνος. Οπότε έχω μόνο μία ερώτηση είπατε πριν στον κύριο Χέγκελ ότι προτιμάτε το αμερικανικό σύστημα. Και από ό,τι κατάλαβα εννοείται τα πρότυπα που έχουν νομοθετηθεί. Ένας, ένας περιβαλλοντικός ε, φορέας το καθορίζει αυτό το, το επίπεδο και κατόπιν το σχολιάζει, το κρίνει η βιομηχανία. Στην Ευρώπη θεωρώ ότι δεν το κάνουμε κάπως έτσι και γι' αυτό και πιστεύω ότι δεν τηρούνται τα δικά μας πρότυπα. Ας είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το να νομοθετούμε και κατόπιν η νομοθεσία να βγει στον κάθε να χρήσουμε. Δεν ισχύει αυτό. Κυρία Κονιέτσινα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που ήρθατε επομένως εδώ να μας μιλήσετε στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι ε, επαναλαμβάνω που δεν υπήρξε ένα πρόβλημα τεχνικό. Ε, είπα ευχαριστούμε που ήρθατε να προσθέσετε στην Επιτροπή μας να μας μιλήσετε και εμείς στα επίσημα τσεχικά κείμενα αναφέρεται ότι έχουμε τώρα κάποια οχήματα ε, τα οποία εσεί παράγετε και έχουν τις μικρότερες εκπομπές της ε, αγοράς και ότι ο ομιλός σας ε, κατέβασε το επίπεδο κατά 14% στα 2 γραμμάρια ανά 100 χιλιόμετρα πρόκειται για τον στόχο του 2015. Αυτά Λες το επίσημο κείμενο όπως το παρουσιάζετε εσείς ως όμιλος. Ισχύει αυτό σήμερα. What I, what I can tell you is that... Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τη διαφήμιση του κ. Βέστερ θα πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός για το τι ανακοινώνει. όσον αφορά το στόλο μας και τις εκπομπές του διοξιδίου, εμείς είμαστε πρωτοπόροι, εν πάση περιπτώσει με άλλες δύο-τρεις εταιρείε στην Ευρώπη. Ήμασταν και είμαστε ακόμα. Δεν είναι πρόκειτο να λέμε τέτοια πράγματα στη διαφήμιση όσον αφορά την κατανάλωση. Όχι, δεν θα λέγαμε ποτέ ότι είμαστε εμεί και μόνοι οι καλύτεροι για τι εκπομπέ. Κανεί δεν το λέει αυτό. Το μόνο το οποίο λέμε στι διαφημίσει είναι ότι τα αυτοκίνητά μα, αυτό το λέμε αυτό που πουλούνται, λέμε ότι είτε συμμορφώνεται με το γύρο 5 είτε με το γύρο 6. Όχι, όχι, κανείς δεν αναφέρει τις εκπομπές ε, στα δημιστικά φυλάδια και ούτε και εμείς. Mm. Ναι, αλλά εγώ θα εννοούσα ότι αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιούν οι πολιτές των αυτοκινήτων σας ή στην Τσεχία σας, ε, το γνωστοποιώ. Αυτό χρησιμοποιούν οι πολιτές στην Τσεχία. Οπότε... Τι γίνεται με αυτά τα 22 λεπτά κατά τα οποία πέφτει το επίπεδο των εκπομπών. Αυτό θα έπρεπε ή όχι να αναφέρεται στα φυλάδια προς τον καταναλωτή. Βέστερ. Επαναλαμβάνω. Όταν λέμε ότι έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε εκπομπές και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Καλά, θα κοιτάξω αν ισχύει και για την ε, Τσεχία. Μιλούμε για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μιλούμε για άλλου είδους ε, ρήπαντες όπως ε, τα οξύδια του αζότου κλπ. Λέει ο κύριος Βέστερ. Κονιέτσα. Όμως, τα οχήματα του ομίλου σας εμφανίζουν αυτήν την ιδιοτυπία των 22 λεπτών που πέφτουν τα, οι, οι τιμές και άλλα τινά. Οπότε στη ΣΥΠΑ υπήρξαν αρνητικές κρίσεις και είχε επιβληθεί και κάποια βαριά καμπάνα. Οπότε, τι λέτε, δεν θα έπρεπε να έχουμε παρόμοια τεστ ε, όπως έχουν οι Αμερικανοί και στην Ευρώπη για την ασφάλεια. δεν κατάλαβα ακριβώς σε τι αναφέρεστε, λέει ο κύριος Βέστερ. Σας είπα επανειλημμένα και λυπάμαι που σας ξαναλέω πάλι το ίδιο. Τι όχι, τίποτα, τίποτα δεν πέφτει, τίποτα δεν σβήνει μετά από τα 22 λεπτά. Ό,τι και να ανακάλυψαν οι αρχές. Ξεχάστε το, δεν, δεν, δεν έχει να κάνει με τη δική μας παραγωγή. Όχι κανένα όχημα μετά τα 22 λεπτά λειτουργίας αφού το έχεις γυρίσει το κλειδί δεν σβήνει τίποτα. Όχι, είναι κάτι που αφορά τη μέτρηση. Μάλιστα λέει πρώτος και εντολός τον κύριο Τούρμες. Δηλαδή δεν σβήνεται, τροποποιείται. Το 80 ή 90%. Έχετε ε, και άλλα στοιχεία να μας προσφέρετε ε, αριθμητικά. Πείτε μου ναι ή όχι, 80, 90, όχι. Α, δεν τροποποιείτε 80 ή 90%. Όχι σίγουρα. Είναι μια τάξη μεγέθους δεν μπορώ να σας δώσω. Γιατί εξαρτάται από πλήθος παραμέτρων αυτή. Πάντως σίγουρα δεν γίνεται σε αυτή την τάξη το μέγεθος. Ο κύριος Τόρμες χωρίς μικρόφωνο. Ε, λέτε τροποποιείτε. Οι πραγματικές εκπομπές ε, ε, οξυδίων των αζώτων εκτοξεύονται και ξεφεύγουν από τα νόμιμα. Ο κύριος ε, ε, Ράρη σας παρουσίασε την έκθεση εδώ και με τα όρια. Σας είπα για το σύστημα EcoDrive που έχουμε και πάνω από 100.000 πελάτες από τους οποίους έχουμε συλλέξει στοιχεία ε, στο μεταξύ. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Στούρμες. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ σας κάνω ερώτηση που μπορείτε να μου απαντήσετε καταφατικά ή ανετικά. Με αυτή την τροποποίηση που κάνετε ε, εκτοξεύονται οι ρήποι, ναι ή όχι. Μετά από 22 λεπτά μέχρι τώρα το κάνατε αυτό. Λάθος λέει ο κύριος. Είστε υπέρ των ε, εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες. Μάλιστα, απολύτως. Γιατί, γιατί καλύπτουν καλύτερα την πραγματικότητα. Για ποιο λόγο είστε υπέρ, δηλαδή? Ναι, σήμερα γνωρίζουμε ότι ε, οι προδιαγραφές NDC για τις δοκιμές ε, δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Χωρίς μικρόφωνο πάλι, κύριε Στόρμες. Λέτε λοιπόν ότι εμείς η Fiat χαιρόμαστε για αυτές τις δοκιμές γιατί αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματική επιβάρηση των ανθρώπων που ζουν στα αστικά κέντρα. Τώρα, αν σας έλεγα εγώ ότι ε, υπάρχει στο περιβάλλον του γερμανικού οργανισμού και μπιέ ότι αντί για να αλλάζει τα 7 μετά από 22 λεπτά, αυτό ε, μπορεί να γίνει μετά από 70 λεπτά. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα τεστ, ε, το real drive emissions, ε, διαρκούν μία ώρα. Δηλαδή, στο παρελθόν τι κάνατε, κανονικές δοκιμές, ότι είναι καθαρός ο ατμοσφαιρικός αέρας ε, στο ε, εργαστήριο και ε, δεν δίνεται δεκάρα τσακιστή για το, τη του ατμοσφαιρικού αέρα στο κέντρο των πόλεων και θεωρείται ότι ισχύει εκεί το ίδιο για το ατμοσφαιρικό αέρα. Η Fiat μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι στο μέλλον δεν θα ξανά τα ίδια. Δεν θα κάνετε τέτοιες τροποποίησεις αντί για σβήσιμο. Κάτι που μοιάζει πάρα πολύ με σβήσιμο, αλλά δεν είναι σβήσιμο, είναι τροποποίηση. Δική σα είναι αυτή η ερμηνεία. Και αυθαίρετη. Γιατί είμαστε υπέρ ε, των, δοκιμών ε, σε πραγματική οδήγηση, γιατί έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει η τεχνολογία, εμείς δεν ήμασταν ποτέ κατά. Πάντα ε, συμμετείχαμε ενεργά και ε, πρωτοπόρα και σε συνεννόηση. Διακόπτει ο κύριος Τούρμες και ρωτάει. Εδώ μπορείτε να μας πείτε με το χέρι στην καρδιά και κοιτώντας μας τα μάτια ότι οι κινητήρες Euro 6 της Fiat τώρα δεν είναι ε, ρυθμισμένες έτσι ώστε μετά από 70 λεπτά να ε, κάνετε τα, τα τεχνάσματα που κάνατε μέχρι τώρα γιατί 60 λεπτά λειτουργεί η διαρκή. Γιατί εμείς έχουμε αυτή την πληροφόρηση και αν ισχύει κάτι τέτοιο, τι να το κάνουμε, πάλι μας κοροϊδεύετε. Είναι λάθος η πληροφόρησή σας. Και με το χέρι στην καρδιά και κοιτώντας στα μάτια. Δεν θα το κάνουμε ούτε με την θεσία, γιατί ούτε τώρα σβήνει τίποτα, ούτε στο μέλλον θα σβήνει τίποτα τα αυτοκίνητά μας είναι πλήρως συμμορφωμένα. Άρα μας λέτε ότι τώρα δεν αλλάζετε αυτά ε, μετά από 70 λεπτά για να ε, ε παρακάμψετε, να βραχικυκλώσετε. Modulate το λέτε. Εμείς το λέμε ότι τα σβήνετε. Εμείς λέτε ότι κάπως τροποποιείτε τη λειτουργία. Εντάξει, κύριε Τούρμες, λέει πρόεδρο, το καταλάβαμε. Ε, ξέρουμε τι ρωτάτε. Όχι, γιατί οι Αμερικανικές αρχές μας προειδοποίησαν ότι για συνθήκες πραγματικής οδήγησης και εκεί χωράει τεχνάσματα και τρίκ. Και τώρα αυτό θα ήταν επιβεβαίωση. Ich weiß nicht genau, was Sie von mir hören möchten. Δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε από μένα. Νομίζω ότι απάντησα, έλαβα θέση για όλα όσα με ρωτήσατε. όσο, ε, όσο, τόσα τεχνάσματα, όσα κάνουμε σήμερα, λίγα τεχνάσματα καθόλου, και το λέω για μας, για τους άλλους δεν ξέρω τι κάνουν, το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Νομίζω ότι σας απάντησα. Και γιατί είμαστε υπέρ πιο λεπτομερών ε, προδιαγραφών που να αποκλείουν κάθε περιθώριο παρερμηνίας και ερμηνείας. Και εδώ δεν είναι σημεολογία το αν σβήνω ή τροποποιώ, υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, δεν αποκλείεται αυτό που ε, ισχυρίζομαι. Το αποκλείω το αυτό που λέτε. Το αποκλείω. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' χαίρομαι που μας κάνετε αυτή την εισήγηση και γιατί αποφάσισε ο Όμιλος να επενδύσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχουμε αυτή την ανακοίνωση τύπου ε, του κύριου Μαρκιόνη και οπότε αυτό είναι πάρα πολύ φρέσκα νέα. Αλλά τώρα για να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την τελευταία έκθεση του Ιταλικού Υπουργείου Μεταφορών. Αφορά επτά οχήματα της ε, Fiat που είναι αντικείμενο εκείνης της ε, έρευνας σε σχέση με το σκάνδαλο. Αυτά δοκιμάστηκαν ε, ή στα δικά σας εργαστήρια και έχουμε την εσωτερική τεχνική υπηρεσία που είναι εκείνη ακριβώς που έκανε τα τεστ και που απέσπασε ε, την έγκριση τύπου από τις Ιταλικές αρχές. Ναι, η ίδια εργαστήρια, οι ίδιοι τεχνικοί. Βέβαια, αυτή η διαδικασία ίδια τεχνική. βεβαια αυτη εκείνους που έκαναν τα τεστ ε, ακολουθούν αυτά τα πρότυπα που ισχύουν για όλους και γενικώ. Ε, έχετε λάβει ιδιαίτερες συγκεκριμένες ε, οδηγίες για το τι πρωτόκολλα δοκιμών θα ακολουθήσετε. Πέστε μας έτσι ε, ενδεικτικά και σύντομα. Ο κύκλος των δοκιμών του αυτοκινήτου είναι σύμφωνα με τους κανόνες και αυτό ε, παληθεύεται. Εύη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί οι Ιταλικές ε, αρχές απευθύνθηκαν στις τεχνικές υπηρεσίες του ομίλου σας, γιατί δεν είχαν τα εκατομμύρια για να επενδύσουν για δικά τους εργαστήρια. Πολύ ωραία λέει κύριε. Επίσης εξηγήστε μου γιατί όλα τα αυτοκίνητα του ομίλου σας που είχαν αυτές τις χείριστες επιδόσεις όσον αφορά τις εκπομπές του, των οξυδίων ε, του αζότου στην εκκίνηση με μηχανή κρύα πολλοί μας είπαν ότι για συγκεκριμένου λόγους συνέβη αυτό ότι είχαν δηλαδή περισσότερες χρήματα σε αυτά τα αυτοκίνητα δεύτερο το εξήγησα και προηγουμένως ότι έτσι όπω είναι τώρα τα πράγματα, κάθε μέρα κάτι προκύπτει. Κάποια εφημερίδα, ένα περιοδικό, κάτι λέει και προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι από πού από πού τα βρίσκουν αυτά, πού παίρνουν τα αυτοκίνητα. Και πολλε φορε δεν είναι ούτε σαφές, ούτε αληθε ότι τα οχήματά μα ε, είναι ε, εκείνα τα οποία είναι τα πιο επιλήψιμα, ας πούμε, αυτά που αξίζουν τις περισσότερες επικρίσεις. Α, μάλιστα, ευχαριστώ. Μπορείτε να μου πείτε ποιος απεφάσισε τα οχήματα του ομίλου σας να μην περάσουν από τα τεστ του Άρτεμις όπως έγινε με άλλα αυτοκίνητα. Για ποιον κύκλο. Urban Artemis. Διευκρινίζει τον κύριο Βέστερη, κυρία Εύη. Διότι. Πού είναι. Α, στην έκθεση αναφέρει αυτόν τον κύκλο δοκιμών Driving Cycle Artemis. Καλά τα πούμε μετά για τις λεπτομέρειες. Πέστε μας για ποιο λόγο. Μετά μια πρώτη δοκιμή για τις εκπομπές για το NDC σε θερμή και κρύα εκκίνηση έχουμε ε, κάποια αποτελέσματα που εξαφανίζονται για τη Λάντζια, για την Τζουλιέτα, ε, Ήψιλον, τη Λάντζια Ήψιλον, συγγνώμη, τη Τζουλιέτα και άλλο ένα μοντέλο. Και στην Ιταλική έκθεση, εδώ στο 7, στο, σχήμα 7, λέει για όλα τα οχήματα τα οποία ε, πέρασαν από αυτή την έρευνα και έχουν τις τιμές αναφοράς. Και κατόπιν στην, ε, στην έρευνα αυτά ξαφανίζουν τα στοιχεία. Γιατί? Δεν ξέρω αν, αν είχαν υπόψη αυτοί που έφτιαξαν την έκθεση αυτά τα στοιχεία. Όχι, όχι, δεν εξαφανίστηκαν τα οχήματα ή τα στοιχεία τους, αλλά ε, παρέσχουμε έγγραφες απαντήσεις κάποια στιγμή. Εκεί ήταν. Κύριε Εύη, πέρασε το πεντάλεπτο και τον λόγο έχει ο κύριος Μποργέζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που είχα την καλοσύνη να έρθετε και ξεκινώ με την εξή ερώτηση. Στην απάντησή σας μου φαίνεται ότι κάπως υπεκφύγατε για να συγκεντρωθούμε σε κάτι το οποίο αφορά την έναρξη της διαδικασίας δοκιμών της ε, Fiat. Δηλαδή το input των δεδομένων όταν γίνονται οι δοκιμές για τις εκπομπές. Δηλαδή, ποιες είναι οι τεχνικές προδιαγραφές που έχετε δώσει προς τους προμηθευτά σας για αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και για θέμα διαφάνειας. Ποιες είναι οι διαδικασίες που είπατε να ακολουθούν οι προμηθευτές. Βέστερ. Τα απαντήσαμε αυτά και εγγράφως. Αυτό το οποίο σίγουρα ισχύει είναι ότι σήμερα έχουμε τρει, τέσσερις, πέντε προμηθευτές οι οποίοι είναι θέση να ε, μας δώσουν αυτά τα συστήματα. Τα συστήματα της ε, εκ των επεξεργασίας των ε, καταλυτών και για όλα αυτά συνεργαζόμαστε με τους ίδιους προμηθευτές. Και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν διαφέρουν. Ας πούμε, ε, τι γίνεται με το φίλτρο για τα σωματίδια κλπ. Και τα, τα διάφορα τμήματα αυτού του καταλήτη, τα διάφορα κομμάτια. Ξαρτάται από το ποιο, για ποιο όχημα μιλάμε, για το τι κυβικά έχει ο κινητήρας. Αλλά γενικώ χρησιμοποιούμε τις ίδιες προδιαγραφές και τους ε, ίδιους προμηθευτές. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο κάνει μετά, κάτι που μας καρεύει μετά η Θα μπορούσατε να μας παράσχετε για λόγους διαφάνειας ε, ένα αντίγραφο της σύμβασης μεταξύ Fiat και της Μανιέτη Μαρέλη για να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι καθημερινές γραμμές που δίνεται γιατί αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό λέει ο κύριος Μπαρκίζου για να μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση τα περισσότερα από τα συμβόλαια τα οποία συνάπτουμε αφορούν τα αυτοκίνητα ε, τα οποία είναι στη διαδικασία παραγωγής και όχι τα πρωτότυπα. Και είναι προς συμφέρον περισσότερο εκείνων παρά ημών το ότι υπάρχουν κάποιες ε, συμφωνίες που διέπονται από το απόρριτο. Υποχρέωση μύθια Κύριε Μπορκέτζη, αν μπορέσετε, λέει πρόεδρος, κάνετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση εγγράφος και θα τη διαβιβάσουμε και θα δούμε τι μπορεί να απαντήσει. Καλά, καλά, θα σας το, το πω και εγγράφος. Αλλά ε, τι γίνεται, οι μηχανικοί δεν μπορούν να μας, να μας δώσουν αυτό το έγγραφο που αφορά αυτό το σημαντικό σημείο γιατί νομίζω ότι αναφερόμαστε στα πρωτότυπα επί των οποίων το πτώσμα των δοκιμών είναι γνωστά σε όλους. Και αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στις συμβάσεις με την Μανιέτη Μαρέλη που αφορούν αυτά τα τεστ. Γι' αυτό επιμένω. Δέστε. Ε, βεβαίως και όπως είπε η πρόεδρος να σας απαντήσουμε αργότερα. Εγγράφος, μετά την ακρόαση. Ναι, αλλά επέβαλα την ερώτηση και ήταν γενικόλογη απάντηση. Για πετε μας ποιες είναι οι αλλαγές που γίνονται σε αυτά τα ίδια αυτοκίνητα όσον αφορά αυτά τα διάφορα προγράμματα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη αλλά και στη ΣΥΠΑ. Πρόκειται για κάποιες τροποποίησεις των αυτοκινήτων που πάνε στη ΣΥΠΑ σε σχέση με αυτό που πάνε στην Ευρώπη. Στη ΣΥΠΑ είπαμε και επαναλάβαμε ότι είναι πιο αυστηρή η έλεγχη, οι προδιαγραφές. Όχι, δεν σε ποια είναι η διαφορά. Λέω ποιες είναι οι αλλαγέ που κάνετε σε σχέση με ε, τους μεν και σχέση με τους δε. Καλά, να σας απαντήσω εγγραφο γιατί είναι πολύ περίπλοκο, απαντά ο κύριος Βέστερ, πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος γύρος. Συνάδελφοι, υποσχέθηκα στους προσκεκλημένους μας ότι δεν θα χάσουν το αεροπλάνο τους. Και θέλουμε να τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση. Τα τρία λεπτά είναι το πολύ, όχι το ελάχιστο που έχετε στη διάθεσή σας. 40 δεύτερα η ερώτηση λοιπόν για να απαντήσει. Ο κύριος Σαλίν. La prima domanda eh, il... Eh, το πρώτο ερώτημα αφορά τις επιπτώσεις όσον αφορά τη βιομηχανία αλλά και την κοινωνία. Και είμαστε να γνωρίζουμε ότι ότι ο περισσότερο κόσμο δεν διαλέγει αυτοκίνητο επί τη βάση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, επί τη βάση τη τιμής. Εσείς θεωρείτε ότι όλα αυτά πρόκειται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αγορά των μικρών διζελοκινητήρων. Σίγουρα ναι. Έχουμε ένα μικρό ε, πάντα, μια μεριά με διζελοκινητήρα και ένα η τέχνη δεν έχει αρντή, βέβαια αν είναι το, η αύξηση του κόστους είναι σημαντική, ε, τότε αυτό δεν είναι εμπορική πολιτική. Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ. Οπότε σίγουρα και θα υπάρχει επίπτωση στην αγορά γι' αυτό. Μάλιστα, θεωρείτε ότι αυτή η αλλαγή για το σύνολο των αυτοκινήτων από τη βιομηχανία πρόκειται να έχει επιπτώσεις ε, για την απασχόληση, δηλαδή για αυτούς που εργάζονται στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Βέστερε, βέβαια, ξέρετε τι λένε όσον αφορά τα υβριδικά, όσον αφορά τα, τους ηλεκτροκινητήρες. Και τι ισχύει σε σχέση με τις εκπομπές. Τι να κάνουμε, να δαπανίσουμε δισεκατομμύρια και μετά όπως έγινε στις ΕΙΠΑ να μην θέλει κανένας ε, το ε, ηλεκτρικό αυτό 500 γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό. Ναι, αλλά τι λέτε όσον αφορά τις εκπομπές. Οι εκπομπές του διοξιδίου θα έχουν επιπτώσεις στους ηλεκτροκινητήρες. Ε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα Και εγώ έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον ηλεκτροκινητήρα. Όχι όσον αφορά τις επιπτώσεις τοπικά, αλλά όσον αφορά το παγκόσμιο αποτύπωμα. Είναι πρόβλημα της μπαταρίας. Και το 2000 είχαμε 10.000 τεραβάτσαν παραγωγή ηλεκτρισμού και η πρωτογενής ενέργεια για να φτιάξουμε αυτό αυτό το ηλεκτρικό φορτίο στην ηλεκτρική ενέργεια ε, χρησιμοποίησε 64-65% μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειες Και Στη συνέχεια πήγαμε στο 25%. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα χειροτέρεψαν. Πήγαμε στο 60% χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι μπαταρίες, αυτή η ηλεκτρική, ε, αυτή η ηλεκτρική ενέργεια. Ε, Εξαρτώμεθα πάρα πολύ από το πετρέλαιο, από τον άνθρακα και γι' αυτό λέω ότι θα είναι επιπτώσεις πάρα πολύ αρνητικές για το παγκόσμιο αποτύπωμα. Είπατε ότι για τα οχήματα Euro 6 αλλάξατε τις τεχνικές ρυθμίσεις για να συμμορφωθείτε με τα πρότυπα για τους δρύπους. Μας είπατε το κάνατε για να προστατευτεί ο κινητήρας. Δεν μπορούσαν γι' αυτό το λόγο να λειτουργούν πάντα τα συστήματα Τώρα τι άλλαξε από το Φεβρουάριο που με το νέο σύστημα και συμμορφώνεστε με τα πρότυπα για τα οξύδια του αζότου και προστατεύετε τον κινητήρα ταυτόχρονα. Τι άλλαξε. Προσπάθησα στην αρχή να το εξηγήσω αυτό όταν μίλησα για τη λειτουργία EcoDrive. Ε, καταγράφονται εκεί τα στοιχεία της οδήγησης και ε, κυρίως στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη από 100.000 οδηγούς ε, έχουμε λεπτομερή στοιχεία πώς χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο και διαπιστώνουμε ότι σχεδόν 95% είναι ε, ταξίδια κάτω από, ε, είναι αποστάσεις κάτω από 60 λεπτά. Κατά μέσο όρο, λοιπόν, φτάνουν σε ένα ορισμένο όριο οι εκπομπές και έτσι έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρες ενδείξεις ε, σε, σε σχέση με το που, σε ποια σημεία μπορούμε να φτάσουμε σε ανώτερα όρια στις ε, τεχνικές ρυθμίσεις, γιατί προσπαθούσαμε να αποφύγουμε κινδύνους που ουσιαστικά είναι ανύπαρκτοι. Προκύπτει από τα στοιχεία. Μάλιστα, λέει η κυρία Μπονιφά, γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα, γιατί αυτή περιπτώσει Και οι προμηθευτές Μπος ε, και Μαγκέτη Μαρέλη από τη μία και εσείς από την άλλη. Ε, ε, πώς κατανοείτε τις ευθύνες, ποιος φέρει την ευθύνη τελικά. Πρόκειται μόνο για τεχνικές ρυθμίσεις, ε, είπαμε, ε, για να προστατεύουμε ταυτόχρονα τον κινητήρα, αλλά και να κάνουμε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για να συμφωνόμαστε με τα πρότυπα. Ε, απάντηση για το θέμα της ευθύνη, το βλέπετε στις γραπτές απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η διαδικασία και δεν θέλω να προσθέσω τίποτα παραπάνω σχέση με τα γραπτά στοιχεία που σας έστειλα, γιατί δεν το κάναμε εξ αρχής, γιατί δεν είχαμε αρκετά οχήματα στην αγορά από το Euro 6 και δεν είχαμε και αυτά τα στοιχεία των οδηγών. Ε, δεν ήταν αρκετά αντιπροσωπευτικό το δείγμα των πελατών για να μπορέσουμε να ε, ρυθμίσουμε λεπτομερέστερα τα οχήματα και να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ από πλευρά μου που ήρθατε σήμερα. Λέει ο κύριο Σούλτσε, μια ερώτηση έχω στην απάντησή σα παριθμών 2. Μιλώ για το γραπτό ερωτηματολόγιο. Πώς αντιλαμβάνομαι μια πρόταση που γράφετε εδώ. Λέτε και ισχυρίζεστε ότι τα οχήματά σας δεν αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται σε δοκιμή. Σωστά το κατάλαβα. Α, μάλιστα, απολύτως. Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται. Δεν το χρειαζόμαστε εμείς για να τις τεχνικές ρυθμίσεις. Καλά, τότε δεν συζητάμε για το ίδιο πράγμα. Ακόμα και η εταιρεία Bosch που ήρθε εδώ μας είπε ότι είναι απολύτω απαραίτητα τα οχήματα να αναγνωρίζουν ότι βρίσκονται στο εργαστήριο και ελέγχονται, έτσι ώστε ε, να ρυθμίζουν αντίστοιχα και το σύστημα ε, ABS για το προκάρισμα των φρένων. Τώρα μας δείτε το αντίθετο. Τι κάνουμε, παράλληλη συζήτηση κοφών. Όχι, όχι. Εμείς μιλάμε για έλεγχο καψέριων και ε, εάν το σύστημα ελέγχου ρήπων ε, ε, ξέρει ότι δοκιμάζεται. Όχι. Υπάρχουν άλλα συστήματα που ελέγχονται ε, που πρέπει να τα γνωρίζουν και που συνεννοούνται μεταξύ τους σε υψηλή ταχύτητα. Εγώ ρώτησα αν το αυτοκίνητο αναγνωρίζει ε, ότι είναι διαδικασία ελέγχου. Δεν ρώτησα αν το σύστημα ελέγχου το ρήπον αναγνωρίζει, αν το όχημα το αναγνωρίζει. Και πόσο σημαντική είναι για σας η ε, γερμανική αγορά. Εξ όσων γνωρίζω, 3 εκατομμύρια από 13. Απαντάει αυτό. Ε, είναι αρκετά σημαντικό, γιατί είπατε ότι δεν σβήνεται μετά από 22 λεπτά. Στη Γερμανία όμως επανειλημμένα αυτό ακούγεται. Γιατί δεν βγαίνετε επιθετικά να κάνετε μια εκστρατεία ενημέρωση ότι είναι λάθος αυτά που διαδίδονται. Διότι, απάντησε. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιδιωτική συζήτηση με τη Γερμανική Υπηρεσία Ελέγχου και έγκριση Οχημάτων. Και γιατί έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην διαδικασία διαμεσολάβησης που έχει αρχίσει. Με την ιστορική μας ε, ε, αρχή έγκριση τύπου, ε, ε, η πρώην Fiat και όμιλος Fiat Chrysler, για όλους τους κινητήρες και για όλα τα οχήματα που παράγονται και πολλούνται είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική είναι υπόκειται σε έγκριση τύπου από το Ιταλικό Υπουργείο Μεταφορών έκαναν την έγκριση του τύπου καλά για τη Μαγνήτη Μαρίλη θέλω να ρωτήσω γι' αυτό σύντομη ερώτηση σήμερα Πώς θα κάνατε την επικοινωνία με το γερμανικό ε, οργανισμό και το Γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών όπως το παρελθόν τους τελευταίους μήνες. Ναι. Πήγαμε γιατί μας κάλεσαν, απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις και παράλληλα είμαστε σε συνεννόηση και με τις Ιταλικές αρμόδιες αρχές που μας είπαν ότι συζητάτε πράγματα που είναι δική μου αρμοδιότητα. Uh, Ευχαριστώ. Στην απάντησή σας ε, στην ερώτηση 8 λέτε για την ευρωπαϊκή αγορά τα περισσότερα ε, Eurocars ε, ή αυτά που παράγονται για την αμερικανική αγορά έχουν λάβει έγκριση τύπου από την Ιταλία. Όμως για αυτά που προορίζονται για την Αμερική και χρησιμοποίησατε την Ολλανδική αρχή. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί. Για ιστορικούς λόγους. Ε, αυτό το έκανε η Chrysler στο παρελθόν. Η FCA είναι συγχώνευση, ξέρετε, της Fiat ε, και του, της Chrysler. Κανείς, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι έκαναν αλλαγές σε σχέση με την έγκριση τύπου. Ε, με, το συμφωνήσαμε με το Υπουργείο Μεταφορών στην Ιταλία και ε, για διάφορους λόγους ε, οι Αμερικανοί την EPA χρησιμοποίησαν και την CARB για τα αμερικανικά και αντίστοιχα για τα ευρωπαϊκά Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία. και λειτουργεί ίσω η διαδικασία. Γνωρίζονται όλοι εδώ και χρόνια, κανείς δεν άλλαξε τίποτα. Μάλιστα, για τον έλεγχο της αγοράς στην Ευρώπη. Για να είναι θεμητή ωραία ανταγωνισμού για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, πιστεύετε ότι αρκεί αυτό το, το υφιστάμενο σύστημα ή χρειάζεται ένα διευρυμένο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε πλήρη συμμόρφωση των οχημάτων. Ξέρετε ότι για τον έλεγχο εκπομπών ε, πρέπει να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργήσουμε τα 160.000 χιλιόμετρα, χρέχουμε τα τέσσερι μόρφωσης. όλα αυτά τα κάνουμε. Το ποσοστό των οχημάτων και τα έγγραφα που που πρέπει να έχετε αν σας ζητηθούν, όλα αυτά τα κάνουμε. Ναι, ναι, εγώ ρωτούσα, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ελέγχουν περισσότερα οχήματα, παραδείγματο χάρη, ε, στο δρόμο, ούτως ώστε οι πελάτες, οι καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στα οχήματα. Απάντηση. Όχι, όχι, ε, πρέπει να φτιάξουμε τους, τους κανονισμούς. Ναι, εντάξει, καλύτερη νομοθεσία. Όμως ε, Φτάνει αυτό. Ε, για να λειτουργήσει το σύστημα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Ε, αρκεί η καλύτερη νομοθεσία να αφήσουμε τους ελέγχους, αυτό μας λέτε. Απάντηση. πρέπει να καλύψουμε αυτά που συζητάμε με καλύτερη νομοθεσία. Έχουμε τη συμμόρφωση στη συνέχεια. Μετά χρειάζονται ανεξάρτητοι οργανισμοί με τις κατάλληλες ε, δεξιότητες για να κάνουν τους ελέγχους. Ο κύριος Νίτερμαγερ, τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, σε σχέση με την απάντηση για το ερώτημα 11. Είπατε το SCR e είναι πολύ ακριβό για μικρά οχήματα. Τι εννοείτε εσείς ε, με μικρά οχήματα, γιατί κάποιοι από τους ανταγωνιστές σας βάζουν στην κατηγορία Β SCR. E Πάντηση. Για το A, πάντα. Και το Fiat, το 500 και για το SCR e υπάρχουν διάφορα είδη SCR e παθητικό που χρησιμοποιήθηκε από κάποιου OEM σε κατασκευαστέ το 2008. Η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων SCR δεν είναι πολύ καλύτερη από έναν καταλήτη αποθήκευση για οξυδία αζότου ή για από ένα ε, RG ε, για υψηλή πίεση, έτσι, για την χαμηλή πίεση αλλάζουν τα πράγματα. Αν πάτε σήμερα στο, αν πάμε στο, από το 2017 και μετά στο RDE, θα πά, πάνε τα παθητικά συστήματα, θα περάσουμε σε συστήματα και το βλέπετε στις ε, αυτές απαντήσεις σε ποιο θα είναι το μέσο κόστος αυτού του συστήματος. Εκτός μικροφώνου. Σύντομα να ρωτήσω. Ε, είσαστε υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας της νομοθεσίας όπως ε, στη ΣΥΠΑ ή υπέρ του τωρινού συστήματος. Τι είπατε, ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Είστε υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας. Η ίδια όρια ουδετεροτητας ιδια ορια εκπομπων ναι, ναι. Τελευταία ερώτηση. Για τις εργαστηριακές δοκιμές, είχαμε κάποιους κατασκευαστές που ρυθμίζανε τα αυτοκίνητα για συνθήκες εργαστηριακές. Δεν μιλάω για τη Fiat. Και δεν ασχολιόντουσαν με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Δεν ισχύει αυτό. Αυτή η παράκαμψη του κύκλου δοκιμών δεν ισχύει. Όλοι συμμορφώνονται με τους κανόνες. Repeating doesn't make it better. Η επανάληψη δεν σημαίνει και βελτίωση. Συμφωνώ απολύτως. Η επανάληψη δεν σημαίνει και βελτίωση. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι αυτός σκοπός, προφανώς. Ένας από τους σκοπούς ήταν φυσικά να έχουμε τις ίδιες συνθήκες για τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων κατασκευαστών. Αλλά το αρχικό κίνητρο για την νομοθεσία αυτή ήταν περιβαλλοντικό και θέμα δημόσιας υγείας. Δηλαδή οι εκπομπές ρήπων να μειωθούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε θέματα ε, αναπνευστικών κυρίως ε, ε, νοσημάτων ή καρδιαγκιακών κτλ. Εσείς τα γνωρίζετε αυτά από τις ε, αποκλίσεις που έχουν οι εργαστηριακές τιμές με τις ε, τιμές σε πραγματική οδήγηση. Χάσαμε το στόχο ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και απέχουμε πόρο. Και τώρα ε, που τα γνωρίζανε αυτά οι εταιρείε και τα επέτρεπαν ή τα επιτρέπουν ακόμα και με διάφορα λογισμικά και τα λοιπά και ρυθμίσεις που δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω χειραγώγηση ε, δεν επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός σκοπός και μάλιστα συνειδητά ε, προκαλούνται ασθένειες, θάνατοι ε, και μενδεχόμεν κίνδυνοι για το περιβάλλον. Γιατρός δεν είμαι, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιου είδους ερωτήσεις. Έχω δει και αριθμούς και μελέτες και εικασίες διάφορες. Το μόνο που μας βοηθάει πραγματικά είναι να ορίσουμε με ακρίβεια τι θέλουμε στο μέλλον και με ποιους όρους και προϋποθέσεις θέλουμε να το πράξουμε. Θυμάμαι μια συζήτηση που έγινε πριν από λίγο που λέει δεν ξέρω να τα γνωρίζετε, πρέπει να το τσεκάρω κι εγώ. Το λέω με επιφύλαξη. Γνωρίζετε όλοι ότι και η κάψη του αερίου Φυσικό αερίου παράγει ε, υψηλέ συγκεντρώσεις οξυδίων του αζότου. Και υπάρχει πηγή αξιόπιστη που ισχυρίζεται ότι όταν έχετε γκάζι στην κουζίνα σας και μαγειρεύετε, ε, παράγεται οξύδιο του αζότου σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από ό,τι στο κέντρο μιας πόλης. Άρα τι εννοείται, ότι βλάπτει το αναπνευστικό, το να μαγειρεύει στο σπίτι σου με γκάζι. Οπότε εντάξει τα αυτοκίνητα και μπορούμε να αγνοήσουμε και να κάνουμε τι θέλουν. Επιπλέον να συνεισφέρει και η κυκλοφορία, δηλαδή δεν φτάνει που έχει τον γκάζι στο σπίτι. Όχι, ο καθένα έχει το μερίδιό του, ο καθένα κάνει τη δουλειά του. Εμεί ασχολούμαστε με τα αυτοκίνητα, με τα άλλα ασχολείται κάποιο άλλο. Απλώ γνωρίζω πολύ λίγα πράγματα σχετικά για να μπορέσω να βγάλω ασφαλή συμπεράσματα για επιπτώσει στην υγεία διαφόρων συγκεντρώσεων αερίων. Μα εγώ ρώτησα για το στόχο της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, πρώτον, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η μείωση εκπομπών ρήπων για λόγους υγείας και για να περιοριστούν οι βλάβες για το περιβάλλον και την υγεία. Εσείς ε, το έχετε δει αυτό ως ε, εργαλείο ρύθμισης αγοράς και μόνο. Η πρόεδρος διακόπτει την κυρία Κάντενμπαχ και δίνει το λόγο στον κύριο Γερμπράντη. Συγγνώμη πρόεδρε, δεν πρόσεχα. Κύριε Βέστερ, ε, παρακαλώ απαντήστε μου με ένα ναι, με ένα όχι. Θεωρείτε το γερμανικό οργανισμό και ε, τον Ολλανδικό που είναι ε, ε, ε, ως ανεξάρτητους οργανισμούς που χαίρουν φήμης, ανεξάρτητοι είναι. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Γκερμπράντη. Και παρόλα αυτά αμφισβητείτε ε, την έκβαση των ερευνών που έγιναν στα αυτοκίνητα ε, Jeep και Fiat. Ε, κοιτάξτε, εγώ είμαι μηχανικός. Για να αποφαθώ πρέπει να έχω στοιχεία. Παραδεχτήκατε τότε στον κύριο Τούρμες ότι μετά από 22 λεπτά το όχημα Fiat ο κινητήρας ε, τροποποιείται και ε, εκπέμπει περισσότερο οξύδιο του αζότου. Έχετε κάνει μελέτες. Εγώ δεν παραδέχτηκα τίποτα. Είπα υπό ε, όρους που δεν γνωρίζω σε λεπτομέρειες κάτι άρχισε να τροποποιείται μετά από 22 λεπτά. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και δεν μπορώ να κάνω εικασίες ή σε ποιο βαθμό συμβαίνει κάτι. Και ήδη έχω αποκρούσει ε, όλους αυτούς τους αριθμούς τους εξωφρενικούς που ακούσαμε προηγουμένως. Α, δεν γνωρίζει Fiat αν το αυτοκίνητό σε αυτό εκπέμπει περισσότερα οξύδια του αζότου όταν τροποποιείται μετά από 22 λεπτά. Εγώ απαντώ στους παραγράφους 5.1 και 5.2, χωρίς μικρόφωνο κύριε Σκευράντη. Ε, η Fiat τα γνωρίζει αυτά. Μα οι πάντες γνωρίζουν και εσείς. Ε, οι πάντε γνωρίζουν ότι άλλο είναι η πραγματική οδήγηση και η δοκιμή στο εργαστήριο. Δεν ρωτάω αυτό, λέει ο κύριο Γκερμπράντη. Μπορείτε να μα πείτε αν γνωρίζει η Fiat εάν τα αυτοκίνητα αυτά εκπέμπουν περισσότερα οξύδια του αζότου μετά από 22 λεπτά όταν τροποποιείται κάπω η λειτουργία του. Εκπέμπει περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να σας πω αν εκπέμπει πάνω από τα όρια. Ναι, εκπέμπει ναι ή περισσότερο οξύδιο του αζότου. Ναι, περισσότερο ναι, αλλά εντός των ορίων παραμένει. Ποιον ορίων. Των νομίμων. Μα, μετά από τα 20 λεπτά δεν υπάρχει νόμιμο λεπτό. Τα νόμιμα λήγουν στα 20. test is only 20 minutes, so if you... Κάθε τεστ ε, δοκιμή για, για αυτά είναι στα 20 λεπτά. Μετά από το 22 δεν υπάρχει νόμιμο όριο, αφού αυτό αφορά τα 20 λεπτά. Πώς το ερμηνεύετε αυτό εσείς με τη νομιμότητα. Μα δεν μιλάω ισπανικά, αραβικά, αγγλικά μιλάω. I uh, Μα σας απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν απαντήσατε, λέει ο κ. Γερμπράντη. Και άλλη ερώτηση. Είπατε ότι έχετε επηρεάσει τη διαδικασία μέσω της ΑΣΕΑ. Αλλά η ΦΙΑΤ συχνά συμμετέχει ε, στην Ιταλική αντιπροσωπεία, σε τεχνικές ομάδες και αλλού. Συμφωνείτε με αυτό. Είναι γεγονός αυτό. Τι να συμφωνώ. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα όπου η ΦΙΑΤ συμμετέχει ως επίσημο τμήμα της Ιταλικής αντιπροσωπείας, γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την έρευνα που κάνουμε εδώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, υπερεύει το όριο πριν, το θα χρησιμοποιήσω λίγο το χρόνο. Μία από τι απαντήσει είχαμε μόνο 12 εκεί. Και ο κ. Σαλήνη μα είπατε όσον αφορά κάποιου είδου εκούσιε βελτιώσει που ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2016 και ότι η Fiat αυτά τα έχει υλοποιήσει. Θέλετε να μας πείτε ε, σε σχέση με αυτό ή να μας ε, πείτε ακριβώ ακριβώς τι, είδου είδους βελτιώσει βελτιώσεις έχετε επιφέρει. Δεύτερο, όπως είπα προηγουμένω όσον ε, αφορά το feedback το οποίο είχαμε από 100.000 ε, και ε, ιδιοκτητών αυτοκινήτων Euro 6 τι γίνεται, πόση, πόση ώρα οδηγάνε, πόσο οδηγάνε κλπ. κλπ. Είδαμε και εφαρμόσαμε το τι είδους ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και έτσι προχωρήσαμε σε βελτίωση σημαντική. Λέει ο κύριος Βέστερ. Και αυτό θα μπορούσε να επιφέρει περισσότερη ε, συμμόρφωση με αυτά στα συμπέρασμα στο οποίο οδήγησε το RDE Βέστερ. Όλες αυτές οι προσαρμογές και οι βελτιώσεις αφορούν την συμμόρφωση με τον κύκλο δοκιμών RDE. Κυρία Κονιέσνα λέει η πρόεδρος. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, γιατί όλα τα κάνατε στρογγυλά, όλα τα κάνατε τέλεια. όσοι είπαν ότι κάτι πήγε στραβό, είπαν ότι δεν τα απολύξαν σωστά ή ότι κάνουν λάθος. Έχετε επίγνωση του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση όσον αφορά ε, τα ελεγκτικά όργανα των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν τα κάνατε σωστά τα πράγματα και δεν υπάρχει ίχνος αμφιβολία σχετικά με αυτά. Εσείς δεν αμφιβάλλετε. Βέστερ. Καθόλου, καθόλου. Αλλά συζητήσαμε για συμμόρφωση προς τον νόμο. Στην αρχή δε σας ανέφερα ότι 100% συμφωνούμε με την πρωτοβουλία βελτίωσης του κύκλου δοκιμών, βελτίωση της νομοθεσίας και την παρέκταση του πεδίου εφαρμογή των εφαρμοστικών κανονισμών ε, και ότι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε σχέση με το τι περιμένουμε. Κονιέσνα. Ναι, αλλά μας ε, είπατε για συνεργασία με τις ΕΙΠΑ και ότι λάβατε υπόψη ε, ε τις πιο αυτές διατάξεις των ΕΠΑ κλπ. Άρα, το ερώτημα είναι γιατί ο όμιλός σας δεν προέβη σε συμμόρφωση ακριβώς προς αυτές τις αυστηρές αμερικανικές διατάξεις όπως ε, επιβάλλει το, το συμφέρον του καταναλωτή. Δεν θα έπρεπε να έχουμε και εδώ κανόνες σαν τους Αμερικανικούς και όλα αυτά θα είχαν επιληθεί. Ήδη σας προανέφερα, λέει ο κύριος Βέστερ, ότι είμαστε υπέρ του να υπάρχει ρύθμιση και προτυποποίηση παγκοσμίου επίπεδου. Όπως κάνουν οι Αμερικανοί. Και για τους διζελοκινητήρες και, και για τους βενζινοκινητήρες. Σας ξεκαθαρίζω όμως ότι εμείς Και χθες και σήμερα και αύριο θα είμαστε υπέρ η ασδήποτε πρωτοβουλία θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα και για σας και για μας και τους πελάτες μας. Ο κύριος Τούρμες, τελευταία ερώτηση. Στα αγγλικά αυτή τη φορά. Είπατε για το άρθρο 5.1 που ε, ορίζει την κανονική χρήση. Έχετε δίκιο. και θα πρέπει να συμμορφώνονται και οι μελέτες και οι δοκίμες. Και ε, για τα φρένα ε, κάνετε άλλες δοκιμές και στην κανονική οδήγηση είναι αλλιώς. Για τις ζώνες ασφαλείας το ίδιο θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Για τις ζώνες ασφαλείας, τι κάνετε, βελτιστοποίηση στις δοκιμές και στην πραγματικότητα είναι λιγότερο καλές. Το ίδιο ισχύει για τις πόρτες, για κανονική χρήση, για την οδηγία. Για τις πόρτες το ίδιο κάνετε. Άλλο στις δοκιμές και άλλο στην κανονική οδήγηση. Αυτό που είναι απίστευτο είναι ε, το εξής. Έχουμε την κανονική χρήση ε, παντού να αναφέρεται στην ε, νομοθεσία με καλό τρόπο και έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι στην κανονική χρήση και στην κανονική οδήγηση για τους ρήπους ε, γίνεται η δοκιμή στο εργαστήριο και όχι μέσα στην πόλη. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συνειδητά σχεδιάσατε αυτοκίνητα ε, όχι με στόχο να προστατεύεται η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και το έχει κάνει και εμένα αυτό η εταιρεία σας. Αποκρούω και απορρίπτω απολύτως όλα αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Δεν υπάρχουν άρθρα 5.1, 5.2 για τα άλλα εξαρτήματα και ανταλλακτικά που με βάση το ενδιαφέρον, το συμφέρον του ε, καταναλωτή είναι για την ασφαλή λειτουργία. Ποια είναι η ασφαλής λειτουργία. The what do you ε, Τι χρειάζεστε δηλαδή για να προστατεύετε εσείς. Τι θέλετε να προστατεύσετε στο EGR. Γιατί σε καμία από τις δεν απαντήσατε με ακρίβεια. Στο EGR, ας πούμε, ε, ε, NOx, TRAPS, τις παγίδες τι θέλετε, ε, οξυδίου του αζότου, τι θέλετε να προστατεύσετε. Εάν λειτουργούν ε, επαόριστον, μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Ε, μπορεί να εκραγούν, μπορεί να έχουν ε, άλλες λειτουργικές αδυναμίες, μπορεί το, το, το κινούμενο, το όχημα να έχει προβλήματα στην κίνηση και στην απόδοσή του. Ε, μπορεί να μην πιάνει τον γκάζι, μπορεί ένα σωρό πράγματα να συμβούν. Συγγνώμη σας, σταματώ εδώ. Υπάρχουν και ECR και άλλα συστήματα υψηλότερης ποιότητας που χρησιμοποιούν άλλοι κατασκευαστές. Εσείς συνειδητά εσκεμένα στους δικούς σας τύπους, τα μοντέλα σας, αγοράσατε πολύ φτηνά μοντέλα ECR, τα οποία σβήνεται ή τροποποιείται μετά από 22 δεύτερα, λέει ο κύριος Τούρμες. Είναι απολύτως ε, λανθασμένο αυτό. Χρησιμοποιούμε τα ίδια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με οποιοδήποτε άλλο ε, κατασκευαστή. Συγγνώμη. Μα δεν είναι η ίδια τεχνολογία. Ορισμένα είναι ε, υψηλότερη ποιότητα και αντέχουν περισσότερο. Αυτή είναι η τελευταία απάντηση. Η απάντηση είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Περίπου τηρήσαμε και το χρόνο μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ήρθατε. Όπως ακούστηκε ήδη, ε, θα γίνουν και άλλες ερωτήσεις ε, ε, για τους συναδέλφους. Προθεσμία για την κατάθεση των επιπλέον γραπτών ερωτήσεων στη ΦΙΑΤ είναι η επόμενη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου. Δικά μας είναι αυτά, κύριε Βέστερ, δεν σας αφορούν, μην σας απασχολούν. Αγαπητοί, πριν φύγετε, σπέστε όλοι να αποχωρήσετε. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε σύντομα. Έχουμε άλλο ένα σημείο στη σε διάταξη και συχνά δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Από τη μία κρούση στην άλλη περνάμε, όπως ξέρετε. Και πρέπει να προετοιμαστούμε για την ανταλλαγή απόψεων. Κάποια στιγμή πρέπει να συζητάμε και τα συμπεράσματα και την έκθεσή μας. Προτείνω τώρα να ακούσουμε ένα σύντομο feedback από τις αποστολές. Θέλω, αν συμφωνούν οι συγητές, να το συνδυάσουμε. Θα κάνω εγώ για το, κοινό κέντρο ερευνών ε, μια εισαγωγή και μετά θα ακούσουμε Ζέλβα και Γκεμπράντι. Όχι ένα λεπτάκι. Ζήτησα να μου πείτε αν συμφωνείτε, αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, 18 και 19 Ιουλίου έγινε η αποστολή. 12 μέλη. Εμείς ε, υποφαινόμενοι και ο κύριος Άλβαμ γι' αυτό. Ε, θα του δώσω το λόγο. Πολύ ε, επικοδομητική η αποστολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε στα εργαστήρια Βέλα στην Ίσπρα. όπου καλύπτουμε τις καλύπτονται οι τεχνολογίες ε, μέτρησης εκπομπών. Επίσης ε, μιλήσαμε για τις εργαστηριακές δοκιμές, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες και τον ε, εξοπλισμό PEMS ε, για τις δοκιμές στον δρόμο. Και εκεί μπροστά στο Ίσπρα κάνα... είδαμε και μια επίδειξη, μια δοκιμή. Μετά κάναμε μια διεξοδική συζήτηση. Είχαμε και αν ε, στις 19 Απριλίου και ακρόαση. Πρέπει να αποφασίσουμε, θα ξανακαλέσουμε στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και πάλι στους εκπροσώπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Με τον κύριο Βλάντι Μυρσούτσα, το διευθυντή, συζητήσαμε με τον κύριο Τζομανίδη Τισάντη και άλλους ε, ειδικού. Προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε όλα τα ζητήματα που είναι σημαντικά για τις δικές μας έρευνες. Ποιος είναι ο ρόλος ε, πρώτα απ' όλα του κοινού κέντρου ερευνών για να καλυφθούν αυτές ε, οι αποκλήσεις τρεις εκπομπών, πώς να χειριστούμε όλα αυτά τα στοιχεία και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε τη, ε, ιστορικά την ανάπτυξη των τεχνολογιών PEMS και RDE για τις νέες δοκιμές δηλαδή και μιλήσαμε για το νέο πλαίσιο, για τη νέα έγκριση τύπου, τη συμβολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών και επειδή υπάρχει μεγάλη... Μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και σε σχέση με αυτά που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό στο οποίο σίγουρα καταλήξαμε και είναι και το μόνο είναι ότι χρειάζεται ένα εξάρτητο οργανισμό με επαρκή πολιτική βούληση για να αντεπεξέλθει στι απαιτήσει των κρατών μελών και ε, να χειρίζεται τι αυτοκινητοβιομηχανίε. Πολύ. Ε, πάρα πολύ υλικό για να τροφοδοτήσει τι συζητήσει μα αλλά και τη δουλειά που κάνουμε σε άλλε επιτροπέ όπω την ΙΜΚΟ παραδείγματο χάρη. Η επίσκεψη και οι συζητήσεις με το Διευθυντή και το προσωπικό μας ε, έδωσαν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τη λειτουργία τη αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια και οι πολλές ιδέες σε σχέση με το πώ μπορούμε στο μέλλον να αλλάξουμε τα πράγματα, να τροποποιήσουμε το σύστημα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζέλμπα και μετά στον κύριο Γκεμπράντη. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, κυρία Πρόεδρε, όπως είπατε προηγουμένως, η Επιτροπή μας ε, και στο Λουξεμβούργο και στη Γερμανία ε, διοργάνωσε ε, αυτές τις αποστολές. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν τα στοιχεία για αυτό το διήμερο από τις 13 Οκτωβρίου και επίσης μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Πολλοί συνάδελφοι και ο κύριος Γκέρμπραντι, συνεισηγητής, συμμετείχαμε στο Φλωράνζ ε, μας υποδέχτηκαν το Γιουμικόρ, οι Εθνικές Αρχές στο Λουξεμβούργο και στο Λάμσχάιμ επίσης στη Γερμανία. Και τους ευχαριστούμε όλους για την ε, φιλοξενία. 21-22 Σεπτεμβρίου έγιναν αυτά. Στο Φλωράζο, όπως σας είπαμε, επισκεφτήκαμε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει καταλήτες. υποδέχτηκε ο καθηγητής Ερμπερτ Λότ, υποδιευθυντής του κέντρου, που μας έδωσε μια συνολική επισκόπηση του Unicorn και τι κάνουν εκεί στην ανάπτυξη και παραγωγή καταλυτών. Παρά τα διάφορα προβλήματα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία από τον κινητήρα Euro 1 μέχρι το Euro 6 είναι πραγματικά success story. και μπορεί να προσαρμοστεί η παραγωγή ε, των κινητήρων Euro 6 και των πετρελοκίνητων. Ε, η νομοθεσία είναι ήδη όριμη ε, και μπορούν να φτάσουν στην αγορά αυτές ε, ε, ε, συσκευές. Ζήτησε εκεί ο διευθυντής που μας υποδέχτηκε περισσότερη δεοντολογία και συμμόρφωση στα όσα ισχύουν. Κάναμε, περιηγηθήκαμε εκεί και το απόγευμα στη συνέχεια πήγαμε και είδαμε τον Υπουργό, την Υπουργό Περιβάλλοντος, την Καρόλ του Λουξεμβούργου και εκπροσώπους του Υπουργείου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υποδομών στο Λουξεμβούργο, καθώς επίσης και το Διευθυντή ε, του Αρμόδιου Οργανισμού SNRC, τον κύριο ε, Κολομουλέχ, ο υπουργό μα είπε ότι το Λουξεμβούργο ενδιαφέρεται πάρα πολύ να λυθεί ε, το πρόβλημα, ενδιαφέρεται πολύ για τι δικές μας εργασίες και τονίζει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη Volkswagen, ε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να έχουμε ε, καθαρό ατμοσφαιρικό αέρα παντού. Χρειάζεται να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, γι' αυτό ζήτησαν ε, και να γίνει μια, ε, ε, ένας έλεγχος από την KPMG στο Λουξεμβούργο για να διαπιστωθεί και τι έχει γίνει όταν εγκρίθηκαν διάφοροι τύποι μοντέλα της Volkswagen. Και υποσχέθηκε ότι θα μας στείλει τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της μελέτης. Η αυτοκινητοβιομηχανία πολλές φορές επιλέγει το Λουξεμβούργο για την έγκριση τύπου, γιατί υπάρχει ένας ειδικός τρόπος με τον οποίο έχει στηθεί το σύστημα ε, και πολλοί ε, βουλευτές εξεπλάγησαν από το γεγονός αυτό παρά το γεγονό ότι το Λουξεμβούργο δεν παράγει αυτοκίνητα, δεν κατασκευάζει αυτοκίνητα, πολλοί κατασκευαστέ επιλέγουν το Λουξεμβούργο να εγκρίνουν τα μοντέλα του. Ε, Στι συζητήσει που είχαμε λοιπόν, ρωτήσαμε διάφορα πράγματα, ιδιαίτερα ε, θέματα. Ε, ε, γιατί δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες και τις αναθέτουν εξωτερικά. Ε, ρωτήσαμε ποιο, το σύστημα έγκρισης τύπου και τι προβλήματα έχουν, ε, πώς έχει υποπτία της αγοράς και επίσης ε, τι γίνεται με τις κυρώσεις και πώς επιβάλλονται. Ο κ. Πολ Φιλίπ από το Υπουργείο Μεταφορών επίσης μας ενημέρωσε. Μετά την παρουσίαση αυτή Ζητήσαμε να μας διευκρινίσουν διάφορα πράγματα νομικά, τι γίνεται σε περίπτωση παραβάσεως, σε περίπτωση defeat devices και, τι είναι, και ποια είναι η νομική βάση για την έγκριση τύπων, ε, για την κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά και τι γίνεται με τις κυρώσεις και πώς επιβάλλονται. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γκέρ Μπράντι για να μας ε, πει τα υπόλοιπα γιατί δυστυχώς δεν ήμουν παρόν σε όλη τη διάρκεια της αποστολής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ συνάδελφε Θάλμπα και κυρία Πρόεδρε ξέρετε πήρε το τρένο για να γυρίσει. Αυτό ήταν πάρα πολύ οικολογικό. Έτσι γύρισε. Και την δεύτερη μέρα. Ε, σε κάποιες ε, εγκαταστάσεις στην ε, Ράινλαντ. Πολύ ενδιαφέρον. Quite interesting to, to... Και εκεί είδαμε τις λεπτομέρειες της παραγωγής. Η διατμόσφαιρα το περιβάλλον των τεστ. Πώς καταρτίζεται. Είδαμε τον ρόλο του οδηγού, θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες κινήσεις ο οδηγός. Υπάρχει μια ε, οθόνη μπροστά. Υπάρχει κάποια καθορισμένη σταθερή ταχύτητα και αν πάει ο ε, ο οδηγός πιο γρήγορα ή πιο αργά, αυτό επηρεάζει τα αποτέλεσματα, οπότε η, η Τουβ είπε ότι... Και Εξαρτάται επομένω από το πώς θα γίνει η δοκιμή για το αν θα υπάρχουν χαμηλότερες ή υψηλότερες εκπομπές. Άρα μπορεί κανείς να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είδαμε πώς γίνεται επομένως το τεστ με τα ίδια μας τα μάτια. Επίσης, μα έδειξαν κάποια PEM που τα είχαν εκεί, πώς αυτά χρησιμοποιήθηκαν ε, κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου δοκιμές αυτός ο κύκλος που κάπως ήταν σαν τον κύκλο δοκιμών RD. Μας είπαν ότι οι εκπομπές με το RD ήταν πέντε φορές ε, πιο υψηλές από ό,τι στο εργαστήριο. Οι λόγοι. Μόνο να υποθέσει μπορεί κανείς την ε, λύση ίσως υπήρχε στον δρόμο περισσότερη επιτάχυνση, ίσως η παγίδα του για το Νόξ δεν ήταν η καλύτερη ποιότητας. Α, και κάτι άλλο που θεώρησα πολύ ενδιαφέρον από πλευράς της επίσκεψης στη Γιούμικορ Υπάρχουν πολλές επικρίσεις όσον αφορά τους παράγοντες συμμόρφωσης. Μας το είπανε έξω από τα δόντια. Ότι δηλαδή η καινοτομία αλλά και σχετικά με τις εκπομπές όλα καθορίζονται μόνο από μία μεταβλητή, την νομοθεσία. Η Κίνα σήμερα έχει θεσπίσει νομοθεσία που είναι πολύ πιο αυστηρή από το Euro 6. Αυτό τι σημαίνει. Φοβούνται ότι η καινοτομία θα μετακινηθεί. Ότι θα έχουν αυτή την καινοτομία εάν εμείς επομένως δεν κάνουμε τίποτα όσον αφορά την νομοθεσία για την παραγωγή αυτοκινήτων. Αυτά ήθελα να σας τονίσω και την πρώτη μέρα. Ε, ευχαριστώ. Εμείς... Και τους δύο. Ε, δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Σαβίνη και Τούρμος, δεν ξέρω κανένας άλλο. Ο κύριος Τζορίνι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μόνο που θα ήθελα να πω ήταν κάτι να συμπληρώσω σε σχέση με το όσα είπαν οι δύο προλαλήσαντες. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής σε σχέση ε, με την Ίσπρα και την επίσκεψη στο κοινό ερευνητικό κέντρο. Είναι πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή για τις εργασίες μας και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο στο τέλος των εργασιών μας να ε, ξαναπάμε ή να τους καλέσουμε ε, για να μας διευκρινίσουν κάποια πράγματα έχει τεχνικές αρμοδιότητες στο κέντρο ερευνών και μάλιστα και δεξιότητες και ε, προσόντα εξαιρετικά. Δεν υπάρχουν ε, προβλήματα τεχνικά περιορισμό. για... Ε, και θέλω να πω ότι υπήρχε και μια πολιτική εντολή που έχει το κέντρο ερευνών στην Ίσπρα Υπάρχουν κάποιες πρακτικές ενδεχομένως εξαπάτησης. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δημοσιεύσεις στα εργαστήρια σε σχέση με τη δυνατότητα ύπαρξης ε, τέτοιας απάτης αναρωτιόμαστε ποια ήταν ε, στη συνέχεια η πολιτική εντολή. Δεν ήταν ε, ε, να γίνουν οι τεχνικές εργασίες για να επιβεβαιώσουμε τις υποψίες ή όχι, γιατί το τεχνολογικό αυτό Ινστιτούτο φυσικά έχει τη δυνατότητα να εξακριβώσει τις πληροφορίες. Όχι, η εντολή ήταν άλλη. Και εγώ ε, σας λέω μόνο αυτά προέκυψαν από την επίσκεψη. Ποια ήταν η εντολή να γίνει ένα βήμα προς τα μπροστά να αναπτυχθούν τα PEMS ε, για να γίνονται οι έλεγχοι σε πραγματικές συνθήκες. Και πραγματικά είναι πολύ καλή η απόφαση. Αλλά γιατί δεν αποφασίστηκαν και τα δύο. Είναι σοβαρότατη αυτή η παράληψη. Γιατί δεν εξακριβώθηκαν αυτά τα στοιχεία, αυτές οι ενδείξεις για απάτη. Αυτή η παράληψη θα πρέπει να καταλογιστεί στους πολιτικούς ηθήνοντες και όχι στους εμπειρογνώμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Και... Ε, φυσικά θα μπορούσε να ε, είχε, μας είχε προειδοποιήσει με πιο αποφασιστικό τρόπο, με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με αυτό που έγινε. Εάν το θέμα συζητήθηκε μόνο ε, στα εργαστήρια και στο νοδικό χάρτη, αντιλαμβανόμαστε ότι λαμβάνοντα υπόψη και το δημόσιο κίνδυνο που αυτό συνιστά και εξαπάτηση των καταναλωτών θα μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα το κοινό κέντρο έρευνα. Πέρα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών υπάρχει μια ασθένεια που μολύνει όλους τους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποποίηση των ευθυνών. Εμείς λοιπόν φέρουμε την ευθύνη στο Κοινοβούλιο να ε, θέσουμε το δάχτυλο τύπου των ύλων και να ε, καταπολεμήσουμε ακριβώς αυτή την τάση. Κανείς δεν θέλει να αναγνωρίσει ότι έχει πλήρη επίγνωση των δεδομένων για να μην χρειαστεί να υπομειστεί την ευθύνη. Η αλλαγή αυτής της νοοτροπίας που είναι επιζήμη για τους καταναλωτές είναι νομίζω αυτό που θα πρέπει να επιδιώξει πάνω από όλα η δική μας ερευνητική επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στούρμες. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπατε για το Λουξεμβούργο. Πολύ ωραία περιγράψατε και την ανταλλαγή ε, απόψεων ε, όταν ήμουν και εγώ παρόν για το κοινό κέντρο ερευνών. Έχει δίκιο ο κύριος Ζωρίνιο. Τα εργαστήρια για τις δοκιμές που έχουν εκεί είναι καταπληκτικά. Άρα, και βέβαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ακόμα καλύτερα στο μέλλον, να αξιοποιούνται καλύτερα. Και λόγος για τον οποίο πιστεύω πρέπει να ξαναφέρουμε τον κύριο Σούτσερ αλλά και τον κύριο Σιμάς και τον νέο διευθυντή, είναι για να δούμε πώς μπορεί το κοινό κέντρο ερευνών να είναι ε, στην καρδιά της εποπτείας της αγοράς και ένα τμήμα αυτού του δικτύου πιστοποίησης εργαστηρίων και έγκρισης τύπων. Πώς μπορούμε λοιπόν να βεβαιωθούμε και να εξασφαλίσουμε ότι οι ε, αναλύσεις και οι πληροφορίες εκεί δεν επηρεάζονται ή δεν ε, μεθερμινεύονται για λόγους πολιτικούς. Πώς θα γίνει αυτό. Χρειαζόμαστε ανεξαρτησία και μια ανεξάρτητη αρχή και πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι είναι ανεξάρτητη από επιρροές. Είναι εξαιρετικό το εργαστήριο. αλλά θα πρέπει με κάποιο ανεξάρτητο τρόπο να λειτουργεί και χωρίς να δέχεται εντολές. Αυτή είναι η ίδια ανάλυση που έχει κάνει και ο κύριος Ζωρίνιο. Όλα τα στοιχεία υπήρχαν, ε, αλλά κανένας δεν τα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που θα όφιλε. Και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε με τον κύριο Σούσκερ και με τον, ε, τον κύριο Σιμάσκη. Αυτή είναι η πρότασή μου. Η πρόεδρος. Αποφασίσαμε ε, να καλέσουμε και πάλι το Κοινό Κέντρο Ερευνών, αλλά θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο, ποιον θα καλέσουμε. Θα το συζητήσουν οι συντονιστές στην επόμενη συνεδρίασή τους. Ας κάνει τις προτάσεις της η κάθε πολιτική ομάδα. Έχει νόημα, είναι λογικό να τους ξαναφωνάξουμε. Και πάλι ε, στα πλαίσια των συζητήσεων που είχαμε για την έγκριση τύπου και την εποπτεία και την επιτήρηση της αγοράς. Πολύ σωστά όλα αυτά. Δεν ξέρω, θέλει κανείς να επανέλθει ή να προσθέσει τίποτα. Όχι. Τελειώσαμε για σήμερα λοιπόν και θα ήθελα να θυμίσω στους συναδελφούς ότι την 5η 20 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 έχουμε πολύ σπουδαία ακροάση με τον κύριο Αλεξάνδρ Ντομπρίντ που είναι ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Μεταφορών ε, στη Γερμανία και με τον ε, Υπουργό των Αρμόδιων από την Κάτω Σαξονία το κρατήδιο. Ε, γεια σας, ραντεβού την Πέμπτη και καλή εβδομάδα.